Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Άρχεται η συνεδρίασή μας. Ηρεμία, ησυχία για να ξεκινήσουμε. Είχαμε μία συνεδρία των συντονιστών που κράτησε λίγο παραπάνω. Η συνεδρίαση πάντως η τωρινή, η συνεδρίασή μας ε, θα είναι μάλλον σύντομη. Υπάρχουν κάποιες ε, ψηφοφορίες οι οποίες μετά και από τη σημερινή συνάντηση του Προεδρείου δεν θα λάβουν χώρα. Έχετε δει την... Ε, μετά από τη διάσκεψη των Προέδρων. Λοιπόν, βλέπετε την ημερήσια διάταξη. Έχετε κάποιες παρατηρήσεις, σχόλια. Alors, j'ai euh, une euh, euh une déclaration à faire aussi une information à donner en ce qui concerne Έχω μια δήλωση να κάνω όσον αφορά δύο κατεξουσιοδότηση πράξεις. Στα αγγλικά. Δύο κατεξουσιοδότηση πράξεις όσον αφορά ε, τα σώματα PPP. Private Public Partnerships Bodies και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις υπηρεσίες τους οργανισμούς λοιπόν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορεί να αντιδράσει εντός δύο μηνών σε αυτές τις κατεξουσιώδεις πράξεις, αλλά δεν μπορούν να υποβληθούν τροπολογίες. Παρακαλώ πολύ, κοινοποιήστε στην ε, γραμματεία μέχρι το τέλος της 18ης Οκτωβρίου εάν προτίθεστε να, ε, ε, να υποβάλλετε οποιαδήποτε ένσταση όσον αφορά αυτές τις δύο κάτι εξουσιοδότηση πράξης. Όσον αφορά τον, το άρθρο 210 υπάρχει επιφύλαξη μελέτης για δύο μήνες. Θα δημοσιευθούν, έχουν δημοσιευθεί μάλλον όλες οι γλωσσικές εκδοχές εκδοχές, τις οποίες θα λάβει το Κοινοβούλιο. Η δίμηνη περίοδος που ανέφερα προηγουμένως μπορεί να επιμηκυνθεί με δύο επιπλέον μήνες. Ε, είναι μικρό το ε, διάστημα δυνατότητας υποβολής ε, αντίρρησης και οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρξει ε, μαζί με την ένσταση και ε, αιτιολογημένη γνωμοδότηση. Και πρέπει να σας πω ότι η προθεσμία λήγει την 25η Οκτωβρίου. Il Όσον αφορά τα συμπεράσματα, θα σας πω δεν υπάρχει, δεν έχουμε ακόμα πρακτικά τουλάχιστον στη διάθεσή μας, δεν, έχουν, δεν έχουμε την εκδοχή αυτή των πρακτικών. Α, έχω και κάτι άλλο να σας πω που το είχα ξεχάσει μετά από αίτημα του εισηγητού. Η έκθεση Ιβάιλο Κάλφιν για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν θα ε, ε, λάβει χώρα σήμερα. Η συζήτηση αυτή θα γίνει την επόμενη φορά. Η οποία επόμενη φορά τελικά θα είναι η 5η Νοεμβρίου. 5η Νοεμβρίου λέω. Θα θυμάστε ίσως ότι είχαμε προβλέψει την ημερομηνία αυτή στη, σαν κανονική συνεδρίαση. Πριν από μερικές εβδομάδες αποφασίσαμε να την ακυρώσουμε τη συνεδρίαση αυτή. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα έχουν λάβει χώρα από χθε μέχρι σήμερα, οι συντονιστές αποφάσισαν ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αυτή η συνεδρίαση της 5ης Νοεμβρίου. Επομένως, σημειώστε το 5 Νοεμβρίου το απόγευμα συνεδρίαση της Επιτροπής Προπολογισμών με σημαντικές ψηφοφορίες. Περνάμε λοιπόν στο κύριο σημείο της σημερινής διάταξής μας που είναι οι διαπραγματεύσεις ε, για τον ε, Διευθυντικό Προϋπολογισμό 2013 και τον τριμερή ε, διάλογο για τον προϋπολογισμό. Θα προσπαθήσω να κάνω μία σύνοψη και θα συμπληρώσουν ό,τι θέλουν οι συντονιστές οι εισηγητές. Έχουμε συζητήσει λοιπόν το ζήτημα του προϋπολογισμού του 2014 ε, και το θέμα των διορθωτικών προϋπολογισμών 2013 καθώς επίσης και για την ε, δέσμη για διαπραγμάτευσης για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Μέχρι τώρα δεν είχε, δεν είχε επιτυχή έκβαση η προσπάθειά μας. Έχουμε ανταλλάξει απόψεις Ωστόσο, εξακολουθούν να ε, υπάρχουν σημαντικά προβλήματα τα οποία δεν έχουν ε, αποσαφινιστεί, δεν έχουν λυθεί και στη διαπραγμάτευση λοιπόν αυτή για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο υπάρχουν αποκλίσεις απόψεις ε, αλλά έχουμε αποκλίσεις απόψεις και για τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς. Ξέρετε ότι στην αρχή της εβδομάδος η Κορεπέρα ενέκρινε το διορθωτικό προϋπολογισμό 8 αυτό το DAB 2, ε, δηλαδή τα 2 δις 900 ε, εκατομμύρια, τα οποία είναι απαραίτητα για να καλυφθούν οι πληρωμές του 2013 και που εξαντλούν το πλαφόν ε, που έχουμε ε, στην διάθεσή μας όσον αφορά ε, τις πιστώσεις πληρωμών για το 2013. Καλό νέο είναι ότι η Κορεπέρ ενέκρινε απαράλλαχτες τις, πρωτο, τις προτάσεις για 2.900.000 αλλά, αλλά έκανε και κάποια σχόλια η Κορεπέρ και στις, ε, στα εκτιμώντας, αλλά και σε μία επιπλέον παράγραφο, συνδέοντας το διορθωτικό προϋπολογισμό 8 με το διορθωτικό ε, προϋπολογισμό 9 καθώς επίσης και με την έγκριση του κανονισμού MFF από το Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο δεν μπόρεσε μέχρι τώρα τουλάχιστον να μου δώσει το αυθεντικό κείμενο το οποίο εκπώνησε η Κορεπέρ. Οι συνεργάτες μας το βρίσκουν λογικό, εγώ όμως το βρίσκω απολύτως παράλογο. Και επιμένω, απολύτως παράλογο. Πρέπει να αποφασίσουμε. Είτε ο προϋπολογισμός είναι μόνο και αποκλειστικά αριθμητικά στοιχεία και επομένως τα σχόλια που μπορεί να κάνει η Κορεπέρε ή το Συμβούλιο των Υπουργών ή το Κοινοβούλιο, μια και το συζητάμε, δεν έχουν καμία νομική υπόσταση και είναι πολιτικά σχόλια και επομένως το γράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια, κάνει το, σχόλιο, το Συμβούλιο ό,τι σχόλια θέλει και το Κοινοβούλιο κάνει και αυτά τα σχόλιά του και κανείς δεν ενδιαφέρεται. We do not mind, λέει ο πρόεδρος στα αγγλικά. Είτε, είτε έχουμε ένα προϋπολογισμό τον οποίο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτός από τα αριθμητικά στοιχεία υπάρχουν και άλλα μη αριθμητικά στοιχεία και επομένως η απόφαση αφορά το σύνολο ε, το οποίο έχει και νομική ε, ε, υπόσταση και από το οποίο προκύπτουν και νομικές δεσμεύσεις και επομένως πρέπει να έχουμε το κείμενο. Εάν έχουμε, όταν λέω έχουμε ένα κείμενο, είτε είναι κανονισμός, είτε είναι οδηγία, το κοινοβούλιο για να ελέγξει το κείμενο αυτό πρέπει να έχει το ίδιο το σώμα του κειμένου στη διάθεσή του. Και εμείς θεωρούμε ότι τα σχόλια, το κείμενο είναι σημαντικά στην προκειμένη περίπτωση. Και πάντοτε έχουμε πει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να είναι συνεκτικό στις δράσεις του και στα λόγια του και επομένως σε όλες τις συνεδριάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, δημόσιου, στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, ε, σε διμερές ε, επίπεδο, σε οποιασδήποτε άλλες συνεδριάσεις, πάντοτε η συμφωνία για το MFF είπαμε ότι είναι δέσμη, το Κοινοβούλιο στο ψήφισμα του της 3ης Ιουλίου ανέφερε σαφώς τις προϋποθέσεις οι οποίες κρίνονται απαραίτητες έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να μπορέσει να κάνει την τελική του ψηφοφορία επί ε, του ε, MFF. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι τρεις και σας τις αναφέρω. Πρώτον, έγκριση χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση των 3,9 δις ε, του διορθωτικού 8. Δεύτερον, ε, η δημιουργία ε, μιας ομάδας υψηλού επίπεδου για να ξεκινήσει τη συζήτηση για την μεταρρύθμιση των ιδίων πόρων και τρίτον, η επαλήθευση ε, ότι δεν υπάρχει πλέον μείζον πολιτικό πρόβλημα ή ε, μείζον πολιτική ε, αντίρρηση όσον αφορά όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία διαπραγματεύτηκε παράλληλα το Κοινοβούλιο. Ξέροντας ότι μονάχα δύο-τρία είναι τα σημεία της διαπραγμάτευσης που μπορούν να προκαλέσουν σημαντικά πολιτικής φύσεως προβλήματα. Εν προχώρησαν και οι διαπραγματεύσεις, αλλά όσον αφορά το κεντρικό μας ζήτημα, τα 3,9 δις του DAB 8, του Διορθωτικού Προϋπολογισμού 8, ε, υπεγράφει σύμβαση μεταξύ του Συμβουλίου και ημών και επομένως δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε ε, ο συνυπογράφων εκ των υστέρων να προσθέσει και άλλη προϋπόθεση. Δεν είναι δυνατόν. Ε, μα μου λένε ξεκινάτε μια διαθεσμική κατά κάποιο τρόπο ε, διαφωνία. Όχι, δεν είναι καθόλου έτσι. Οποιαδήποτε σύμβαση, μια σύμβαση ας πούμε ε, γάμου έχει υπογραφεί και από τους δύο. Δεν μπορείς μια μέρα μετά το γάμο και μετά την υπογραφή της σύμβασης να πεις άξιες κάτι, είχα ξεχάσει κάτι, θέλω να το προσθέσω. Υποχρεούσε να κάνεις και το α ή β ή γ πράγμα συμφωνούμε, υπογράφουμε μια σύμβαση και βεβαίως ε, το είπαμε και εμείς και ο εισηγητή, το είπαμε δημόσια, το είπαμε ιδιωτικά σε όλα τα κράτη-μέλη που τους αφορά το θέμα, το είπαμε και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, μπορούμε να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα και όσο γίνεται με πιο σωστό τρόπο να ε, ε, προχωρήσουμε σε κάποιες, σε, σε κάποιες κινήσεις έτσι ώστε να αποζημιωθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα ε, χώρες οι οποίες υπέστησαν το, την άνοιξη πλημμύρες. Ξέρουμε ότι υπάρχουν καταστάσεις ε, οι οποίες ε, αφορούν φυσικές καταστροφές ή μη προβλέψιμες καταστάσεις και στις οποίες θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις. Το Συμβούλιο σε επίπεδο Υπουργών πρέπει να ψηφίσει έτσι ώστε ε, να ψηφίσει μετά και το Κοινοβούλιο. Το, το Συμβούλιο ψηφίζει πριν από το ε, Κοινοβούλιο. Πριν από τις 30 Οκτωβρίου το νωρίτερο δεν μπορεί να ψηφίσει το Συμβούλιο. Επομένως έχουμε δύο μεγάλες δυσκολίες. Και ένα τρίτο σημείο, το οποίο δεν έχει ρυθμιστεί ακόμα, το οποίο δεν παρουσιάζει τόσο μεγάλο βαθμό δυσκολίας, για την δημιουργία της ε, ομάδας αυτής υψηλού επίπεδου προχωρούν οι διαδικασίες, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διαφωνίες, γιατί ξέρετε συμβαίνει συνήθως όταν ξεκινάμε κάτι καινούριο, είναι όλοι λίγο πιο προσεκτικοί. Επομένως το κλίμα είναι θετικό, υπάρχει και βούληση ε, σύγκλησης απόψεων και βούληση για να επιτευχθεί κάτι σωστό. Αλλά δεν κινούνται οι διαδικασίες τόσο γρήγορα ώστε να είμαστε έγκαιρα έτοιμοι Euh, ε, και επομένως ε, δεν προχωρούμε πολύ. Η Κορεπέρα αφιέρωσε χθες το απόγευμα την απογευματινή ε, συνεδρίασή του σε αυτήν την ομάδα υψηλού επίπεδου, αλλά δεν έχουμε κανένα γραπτό σημείωμα ή υπόμνημα για τις συζητήσεις που έλαβαν χώρα στην Κορεπέρα. Euh, par écrit euh, auprès Γραπτός ενημέρωσα και τον πρόεδρο Σούλτς και τη διάσκεψη των προέδρων για, τον, ε, για την κατάσταση και έχοντας συζητήσει και με τους συζητητές κατέληξα στο συμπέρασμα ότι μπορούμε να κρατήσουμε την ημερομηνία της 23ης Οκτωβρίου σαν ε, ημερομηνία ψήφισης της δέσμης MFF, αλλά αυτό προϋποθέτει ότι η πίεσή μας προς το Συμβούλιο θα είναι πάρα πολύ μεγάλη και ότι δεν θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε τα διάφορα στοιχεία της δέσμης MFF σήμερα, πέμπτη απόγευμα, στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, γιατί δυστυχώς δεν είχαμε το χρόνο να διευθετήσουμε αυτές τις ε, ε, διαφωνίες και επομένως θα γίνει μια έκτακτη συνεδρία στη Δευτέρα απόγευμα. Σήμερα το πρωί η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε να αναβάλει το σύνολο των ψηφοφοριών που σχετίζονται ε, με το MFF. Και ενώ το πι δέλτα πι. Και επομένως στις 19 Οκτωβρίου θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό και αφορά όλες τις ψηφοφορίες ε, ε, ε, και τις νομοθετικές και τις δημοσιονομικές. Και είπαμε ότι στην προκείμενη περίπτωση οι διαφωνίες, είτε πρόκειται για διαφωνίες δημοσιονομικές είτε νομικές, οδήγησαν σε αυτήν την δυσχερή κατάσταση. Θα πρέπει λοιπόν να εξαχθούν τα συμπεράσματα και να δούμε ποιος θα, ποιος θα είναι ο αντίκτυπος αυτών των καταστάσεων. Ε, έχουμε περισσότερο χρόνο λοιπόν να διαπραγματευτούμε και αυτό έχει και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Το μειονέκτημα αφορά την δυνατότητα δημιουργίας αυτής της ομάδας υψηλού επίπεδου, ποια θα είναι η σύστασή του, ποιες διαδικασίες θα ακολουθήσει, ποιος θα προεδρεύσει, ε, ποιο θα είναι το θεματολόγιο του, το χρονοδιάγραμμά του κτλ. Εάν έχουμε ένα μήνα παραπάνω, βεβαίως ε, θα μπορέσουμε να ε, έχουμε και ένα πραγματικό κανονισμό και ένα καταστατικό κτλ. Αυτό ήταν το πλέον έκτημα. Έχουμε όμως και ένα μείον έκτημα θα υπάρξει επικάλυψη με το ετήσιο πρόγραμμα που αφορά τον προϋπολογισμό και επομένως θα επικαλυφθεί, θα επικαλύψει μάλλον κατά κάποιο τρόπο τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του 2014. Στις 23 Οκτωβρίου δεν θα ψηφίσουμε το ΠΔΠ και όλα τα κείμενα που συνδέονται ε, με το ΠΔΠ, αλλά θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες μας για τον προϋπολογισμό έτσι ώστε σύμφωνα και με το αρχικός προβλεπόμενο ε, χρονοδιάγραμμα να είμαστε σε θέση την 14η Νοεμβρίου να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο. Η πρώτη ε, διαμεσολάβηση ε, ξεκινάει ήδη τον επόμενο μήνα. 7 Νοεμβρίου η πρώτη, ο πρώτος τριμερός διάλογος, 11 Νοεμβρίου δεύτερη διαμεσολάβηση και μάλλον η τελευταία γνωρίζοντας ότι η χρονική προθεσμία για την έγκριση προπολογισμού είναι η 13η Νοεμβρίου και επομένως η ψηφοφορία της δέσμης ΠΔΠ θα λάβει χώρα την 19η και επομένως αν έχουμε συμφωνία με το Συμβούλιο σε μία από τις ε, διαμεσολαβήσεις τότε την 19η του μηνός θα έχουμε την τελική έγκριση του προπολογισμού 2014. Πρακτικώς αυτό σημαίνει ότι θα αλλάξουμε διαπραγμάτευση. Θα έχουμε δύο-τρεις δέσμες, δέσμη πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, δέσμη του διορθωτικού προϋπολογισμού υπαριθμών 9 που συνδέεται με, το συνολικό, με τη συνολική καταβολή και μετά τον προϋπολογισμό του 2014. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει ας πούμε δύο-τρεις ε, μικρότερες δέσμες. Τώρα θα έχουμε μία τεράστια δέσμη. Εκ των πραγμάτων λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο ε, και παρότι μιλάμε για προπολογισμού δύο διαφορετικών ετών, η συζήτηση θα γίνει ταυτόχρονα. Επομένως, διαπραγματευόμαστε την εφαρμογή, την υλοποίηση της πολιτικής συμφωνίας για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, πράγμα που σημαίνει ότι θα ψηφιστεί ο κανονισμός ε, ΠΔΠ και η διαθεσμική συμφωνία. Επίσης, ψηφοφορία επί του διορθωτικού προϋπολογισμού υπαριθμών 6, που δεν ε, τον έχουμε ακόμα όμως, τον ε, διορθωτικό προβληματισμό υπορριθμών 7, τον οποίο έχουμε, τον 8, που δεν τον έχουμε. Όλες αυτές οι ψηφοφορίες είναι ε, μαζί με τη δέσμη ΠΔΠ για την 19η του μηνός. Και επίσης θα συζητήσουμε ε, τα, την αποζημίωση για τις, ε, για του, τις πλημμύρες 400 εκατομμύρια ε, και τον πρόσθετο προβληματισμό 900 εκατομμύρια μαζί με το διορθωτικό υπαριθμό 9, μαζί λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ του Συμβούλιο, το, το, το, μεταξύ του Συμβουλίου Κοινοβουλίου Κομισιών σχετικά με τους ε, διαθέσιμους πόρους και σχετικά ε, με τις εγγραφές που αφορούν τις πιστώσεις υποχρεώσεων. Από εκεί και πέρα. Θέλουν οι εισηγητές το λόγο να συμπληρώσουν τίποτα σε αυτά που σας είπα. Ε, well, Chairman, actually this Jan Γένσεν; Μα ε, το προπολογισμό του 2014 βασικά δεν θα ήταν αυτός ο τριμερής διάλογος. Χάνεται όμως μέσα στην ομίχλη όλων αυτών των προβλημάτων με τους, ε, το σχέδιο διορθωτικών προϋπολογισμών και το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ανταλλάξαμε απόψεις για την ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό του 2014 και οι αντιδράσεις από την πλευρά του Συμβουλίου δεν μας εξέπλησαν. Ξαν. Προφανώς δεν συμφωνούν με το γεγονός ότι ψηφίσαμε ένα προπολογισμό ο οποίος υπερβαίνει τη δική τους πρόταση. Και όχι μόνο τη δική τους, αλλά και κατά και την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ιδιαίτερα για το μέσο ευελιξίας. Για τα διαρθρωτικά ταμεία πιστεύουν ότι η σε αυτή πρωτοβουλία για τη νεολαία θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί λέει από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και να βρείτε αλλού τα λεφτά, είπε, να όχι φρέσκο χρήμα. Αλλά έχουμε τη χρηματοδότηση έξτρα για την Κύπρο και για τους απόρους Και ε, το Συμβούλιο λέει και αυτά να τα πάρουμε από το Κοινωνικό Ταμείο. Επίσης, ε, για τις εξωτερικές υποθέσεις, όπου ξεπερνούμε και πάμε στο μέσο ευελιξίας, μας λένε πάλι να τα βρούμε απαλού. Νομίζω ότι ε, η ανθρωπιστική βοήθεια είναι κάτι σημαντικό και ότι θα πρέπει να υπάρχει περισσότερο περιθώριο, ψηλότερο σε κάποιες περιπτώσεις και κατηγορίες. Άρα μάλλον θα μπλέξουμε. Χρειάζεται εκτενή συζήτηση για το τι ψηφίσαμε και πώς ψηφίσαμε. Γιατί έχουμε πολύ ε, ατράνταχτα ε, επιχειρήματα και για τους οργανισμούς. Ας πούμε, πολλοί τρέχουν σημαντικοί σήμερα στη Λαμπεντούζα και τους τάζουν λαγούς με πετραχίλια, ενώ εμείς βάλαμε το χέρι στην τσέπη, 2,5 εκατομμύρια παραπάνω για το Frontex και έξτρα για το Eurosur, ε, για να βοηθήσουμε κάποιους στην Αφρική για να εξηγήσουμε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα στην Ευρώπη όπως τους λένε οι δουλέμποροι. Αυτά ε, είναι θέματα που έχουμε πάρα πολύ ε, γερά επιχειρήματα απέναντι στο Συμβούλιο, αν τα εξηγήσουμε όταν έρθει η ώρα της πραγματικής συζήτησης. Είμαστε έτοιμοι να μπούμε και σε πολύ μεγάλες λεπτομέρειες. Είδατε. Υπάρχουν και ε, διαφορετικά επίπεδα πληρωμών από αυτά που προτείνει το Συμβούλιο. Όχι απλώς επαναφέραμε τα ποσά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι κόκκινη γραμμή. Πιο κάτω δεν πάμε. Αλλά στην ανάληψη υποχρεώσεων έχουμε προσθέσει περισσότερα και δεν θέλουμε να διαγκώσουμε το πρόβλημα της διαφοράς μεταξύ των υποσχέσεων και των πραγματικών μας πληρωμών. Και σε αυτή την περίπτωση δηλαδή θα χρειαστούν συζητήσεις. Βασικά όμως πρέπει να πω ότι βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση που εξηγήσατε κι εσείς ότι είναι όλο ένα μεγάλο πακέτο, μια μεγάλη συζήτηση. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορώ να το αλλάξω. ούτε μου διευκολύνει τα πράγματα, αλλά νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι η διορθωτική, διορθωτική προπολογισμή του κυρίου Λαβία και όλη αυτή η υπόθεση επίλυσης των προβλημάτων για να ανοίξει ο δρόμος και να δώσουμε και εμείς τη σύμφωνη γνώμη μας για το πολιτισμό συνολικό πλαίσιο. Ευχαριστώ. Ωραία. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι το πολύπη έχει καταλήξει να γίνει θύμα πλημμύρα. Τέλος πάντων. Θα μιλήσουν και οι υπόλοιποι εισηγητές και όλοι όσοι ζητήσουν το λόγο, αλλά θέλω να υποφεληθώ εδώ από την παρουσία του Γενικού Διευθυντή Προϋπολογισμών της Κομισιόν, τον οποίο ευχαριστώ για την παρουσία του, και θα ήθελα να του θέσω ένα ερώτημα που να το σκεφτεί ενώ θα μιλούν οι υπόλοιποι. για αυτά που μόλις είπε η Αν Γένσεν ως προς τις δηλώσεις που γίνονται από την Κομισιόν, από το Συμβούλιο και από τις αρχές του Κοινοβουλίου για τις επιπτώσεις και το νόημα της πρόσφατης τραγωδίας στη Λαμπεντούζα ε, στα ανοιχτά της Μάλτας όπου τίθενται ιδιαίτερα ανθρωπιστικά προβλήματα όπως και από τον εμφύλιο στη Συρία. Όλοι βέβαια συγκινούμαστε ιδιαίτερα από όλα αυτά και χαιρόμαστε γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να κάνει κάτι. Κατανοούμε ότι αυτό σημαίνει βέβαια πληρωμή, πληρωμές. Αλλά λόγω των τεραστίων δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή δημοσιονομικά θα ήταν για μας πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ακριβώς σε ποια θέση και ποιο έτος θα τοποθετηθούν οι δαπάνες αυτές και σε ποια κατηγορία θα μπουν οι προβλέψεις ή οι πληρωμές αυτές. Ευχαριστώ λοιπόν. Ο Τζοβάνι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπε και μόλις η Αν Γένσεν, χθες ο τριμερής διάλογος στην ουσία ήταν μία συγκέντρωση ας πούμε προβλημάτων των διορθωτικών προϋπολογισμών 2013. Ε, Επιτρέψτε μου λοιπόν να κάνω κι εγώ μία μικρή σύνοψη προς τους συναδέλφους και να προσθέσω και μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί έστω και αν ε, ε, συχνά έτσι συζητάμε για κάποια επιμέρους ζητήματα, καλό θα ήταν να έχουμε και μια γενική έποψη για να μπορέσουμε να πάρουμε αποφάσεις. Όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 6 και η σειρά που θα ακολουθήσω δεν είναι ε, ανάλογα με τη σημασία τους, αλλά με, το, με τους αριθμούς τους. Σχέδιο διορθωτικού υπολογισμού 6 λοιπόν είναι σαφές ότι δεν έχει συζητηθεί στο Συμβούλιο, δεν έχει ελεγχθεί από το Συμβούλιο, αφορά τα έσοδα ε, και την αναθεώρηση ε, των ε, εσόδων βάσει του ΑΕΠ. Και εδώ έχουμε να σημειώσουμε μία μείωση των τελωνιακών δασμών. Αλλά βεβαίως θα πρέπει να περιμένουμε και την τελική θέση του Συμβουλίου ο διορθωτικός προπολογισμός 7 που σχετίζεται με το Κοινωνικό Ταμείο 2013 και με το ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ οπωσδήποτε αναφέρεται στις επιπτώσεις σε μια συμφωνία σε επίπεδο συμβουλίου, τότε δηλαδή ε, που επετέφθη συμφωνία για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Πρόκειται λοιπόν ε, για την έκδοση αποζημίωσης για τρεις χώρες, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, ε, με 130 και 20 εκατομμύρια ευρώ. Η επιπλέον, η πρόκειται για επιπλέον κονδύλια, τα οποία όμως συνδέονται με τη συμφωνία ΠΔΠ. Το Κοινοβούλιο θα αξιολογήσει και θα μελετήσει αυτόν τον ε, διορθωτικό προϋπολογισμό όταν ε, θα επιτευχθεί συμφωνία επί του προϋπολογισμού υπαριθμών καθώς επίσης και στα άλλα σημεία τα οποία έχουμε αφήσει σε εκκρεμότητα, διότι σχετίζονται με το δημοσιονομικό πλαίσιο. Όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού, υπαριθμών 8, πέρα από την βούληση η οποία φαίνεται να εμφανίζεται σε επίπεδο κορεπέρ, ε, υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο θέλω να σχολιάσω σε σχέση με την ανάγνωση που έχει κάνει ε, το, η κορεπέρ και ε, προκύπτει ένα ερώτημα ίσονος σημασία εργασίας ε, βέβαια γιατί ε, στην ουσία αναφέρεται σε ένα μικρό ποσό σε σχέση με τα έσοδα και μετά μιλάμε για 14 κάτι ε, δις ευρώ που γνωρίζει πολύ καλά η Κομισιόν ε, ένα ποσό ε, για το οποίο η Κορεπέρ θέλει κάποια λίανση του διορθωτικού προϋπολογισμού υπαριθμών 8. Θα πρέπει να ξέρουμε αυτά τα 14,7 ε, εκατομμύρια με τι συνδέονται εάν έχει υπάρξει εσφαλμένη, ε, αν έχει υπάρξει εσφαλμένος υπολογισμός ε, αποφάσεις που έχουμε πάρει με, τον, ε, ε, με το Ταμείο Λεγγύης, που ακριβώς υπάρχουν τα λάθη κτλ. Τώρα, για το σχέδιο δοχετικού προϋπολογισμού υπαριθμών 9, είναι σαφές ότι η πρόταση τη Κορεπέρη, αν θέλετε καλύτερα η πρόταση του Συμβουλίου να χρησιμοποιηθούν 400 από τα 900 εκατομμύρια για να χρηματοδοτηθεί το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης είναι κάτι που πρέπει να μας οδηγήσει σε σκέψεις. Η μείωση του γενικού ποσού. Θα πρέπει να μας πει η Κομισιόν μέχρι ποιο βαθμό αυτή η μείωση μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδι ή να προκαλέσει επιβράδυνση κάποιων ε, ερευνητικών ε, προγραμμάτων ή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων γενικά. Και εδώ στρέφομαι στην Κομισιόν ε, και ακόμα μια ερώτηση και ζητώ συγγνώμη γιατί έκανα πολλές ερωτήσεις αλλά νομίζω ότι είναι σαφές ότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι περί τίνος πρόκειται και υπάρχουν κάθε τόσο νέα στοιχεία. Κατά την άποψη της Κομισιόν λοιπόν, ποιες είναι οι επιπτώσεις, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις ε, μιας μη ψήφισης του σχεδίου Διευθυντικού προϋπολογισμού υπαριθμών 8 ε, στο, στην ε, Σύνοδο Ολομελία ε, του Οκτωβρίου και η αναβολή, η παραπομπή μάλλον σε, στην συνεδρία, συγγνώμη, στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις, θα υπάρξουν αντίκτυποι στην ταμιακή επάρκεια της Κομισιόν. Ε, και θα υπάρξουν και κάποιες ε, λειτουργικές ε, δυσχέρειες. Ευχαριστώ πολύ την Κομισιόν εκ των Προτέρων για την απάντηση που θα μας δώσει. Ευχαριστούμε Τζοβάνι, ήταν σαφές η Μόνικα. Αγαπητέ Πρόεδρε, για τον προλογισμό του Κοινοβουλίου εγώ τι να πω σε σχέση με όλα αυτά. Ο Τζοβάνι Λαβία ε, τα είπε και θα περιουστώ σε αυτά που ανέφερε για το διορθωτικό προϋπολογισμό. Μετά τη χτεσινή συζήτηση ανέκυψαν πραγματικά και εμφανή προβλήματα. Ε, το βασικό μου ερώτημα εμένα ποιο είναι τελικά. Εμείς ως Κοινοβούλιο έχουμε θέσει μια προτεραιότητα. Ένα κέντρο βάρους, πολλά σε διάφορους τομείς, αλλά είναι ιδιαίτερο που θελήσαμε να πούμε ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποχρηματοδοτείτε. Και αυτό είναι η έρευνα. Μπορεί να έχουμε διάφορους οργανισμούς, ε, επιμέρους, να τα συζητήσουμε σε λεπτομέρειες. Αλλά έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, ένα μεγάλο μπλοκ που είναι η έρευνα. Και σωστά θελήσαμε και για την καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανταγωνιστικότητα κτλ. να θέσουμε προτεραιότητες. Έκανε μια πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή 509 εκατομμύρια συνολική μεταφορά. Ωραία αυτά και καλά. Εμείς τι χρειαζόμαστε. 400 για τους πλημμυροπαθείς, ε, γύρω στα 100 για τη Συρία για να το χαρακτηρίσω έτσι και το, το σύνολο που εντάσσεται εκεί ανθρωπιστική βοήθεια, πρόσφυγες κτλ. 100 εκατομμύρια για το Συριακό γενικά και αν θυμάμαι καλά να τα κοιτάξω λίγο για την έρευνα που ε, χρειάζεται 327-328 εκατομμύρια και πρότεινε περικοπές 3.31. Ε, Το ίτερ έχει καθυστερήσει έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν έχει ε, καθυστερήσει κανένα πρόβλημα. Κάθε χρόνο τα ίδια βλέπουμε με το ίτερ. Του χρόνου δεν θα το γράψουμε στο πίνακα γιατί διανύζεται αυτή η ε, μεταφορά από χώρα σε χώρα και θα έχουμε προβλήματα στο επόμενο PDP ε, ή από το 2016. Ας είναι. Εμένα δεν μου είναι σαφές τι γίνεται στο προπολογισμό του 2013. Ξέρετε ότι έχω μακρά εμπειρία στη γεωργία και σε ε, διαφορά άλλα πράγματα. 55 δισεκατομμύρια έχουμε συνολικά, έτσι δεν είναι. Αν βγάλουμε τα 600 εκατομμύρια που μεταφέραμε για το 2014 ε, για τη γεωργία. Λοιπόν, εάν κάπου μπορούσαμε να βρούμε 200 εκατομμυριάκια, όχι πολλά, για να αποφύγουμε, μάλλον να αυξήσουμε σε 709 τη συνολική μεταφορά και το μεταφέρουμε στην έρευνα, τότε μπορούμε να αφαιρέσουμε πολλές έγνοιες από την Αν για το 2014. Δεν μπορούμε να υποχρηματοδοτούμε την έρευνα. Τα άλλα, τα επιμέρους, τα μικρά, αν θέλετε, μπορούμε να τα συζητήσουμε. Αλλά τέτοια γενική υποχρηματοδότηση της έρευνας δεν επιτρέπεται δεν μπορούμε να τη δεχτούμε. Ήδη το 2014 έχει υποχρηματοδότηση. Ε, για το 2013 είναι 192 σίγουρα αυτά που χρειαζόμαστε, το στρογγυλεύω 200. Σε αυτό το τεράστιο προπολογισμό δεν μπορούμε να βρούμε πουθενά 200 εκατομμύρια. Αλλιώς με πιάνει απογοήτευση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και τελικά το 2014 στην Επιτροπή Κοκομπού πρώην και τώρα κόντε, Επιτροπή Ελέγχου δηλαδή, διαβάζω για το 2013 ότι κάπου περίσσεψε ένα δισεκατομμύριο, ε, θα τραβώ τα μαλλιά μου. Θα εξοργιστώ και ζητώ συγγνώμη που τα λέω έτσι και πρέπει και να φύγω αμέσω, γιατί έχω άλλη ενηλυμένη υποχρέωση. Θα σας παρακαλούσα να λάβετε υπόψη μια μικρή πρόταση που έχω υποβάλει. Αν ισχύουν αυτά που άκουσα, θα μπορούσε το Συμβούλιο μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου να φροντίσει να μας αφαιρέσει αυτές τις έννοιες και τα προβλήματα. Και θα συμφωνήσουμε και με τα ντάπτα τα υπόλοιπα, τους ε, διορθωτικούς προπολογισμού. Ευτυχείς δεν θα είμαστε έτσι κι αλλά με βαριά καριά θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. Ήθελα να το πω, γιατί νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να βρούμε κάπου αυτά τα 200 εκατομμύρια για συνολική μεταφορά για την έρευνα γιατί ξέρω ότι είναι και το Συμβούλιο ευαίσθητο για την έρευνα. Και δεν θα πρέπει να ανοίξουμε μέτωπο τώρα, να εκτεθούμε για το 2014 που θα υπάρχουν έργα τα οποία θα καθυστερήσουν λόγω υποχρηματοδότησης. Και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας για την καινοτομία και τα συναφή. Ευχαριστώ. Je comprends tout à fait, euh, Monica. Ναι, το καταλαβαίνω, Μόνικα, το καταλαβαίνω. Γιούτα Χάουκ, πάρα πολύ σύντομα, για να συμπληρώσω αυτά που είπε η Μόνικα Χόλμαϊερ μόλις. Δεν ισχύει ότι το Συμβούλιο θέλει να ε, ε, φάει τα λεφτά αυτά από τη συνολική μεταφορά ή δεν ισχύει 100%. 14,7 εκατομμύρια που λείπουν και έχουν βάλει χέρι και στην έρευνα στον ΤΑΜΠ 8. Παντού κάνουν περικοπές και στην έρευνα. Βγαίνουν ε, τις Κυριακές στα μπαλκόνια, δεν ξέρω, κάνουν μεγάλες ε, εξαγγελίες και βγάζουν ωραίους λόγους και μετά δίνουν ψίχουλα. Hélas, vous avez raison, l'une et l'autre. Δυστυχώς. Κύριε Γενικέ Διευθυντά, να απαντήσετε, έχετε πολλά θέματα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα. Καταρχήν, για τη Λαμπεντούζα. Ο πρόεδρος Μπαρόσο ανακοίνωσε τις προάλλες, όταν επισκέφθηκε τη Λαμπεντούζα, θα κινητοποιήσει 10 εκατομμύρια ευρώ. 18. Ε, Που θα, όπου θα γίνει μια μεταφορά στα πλαίσια του προϋπολογισμού και 14 εκατομμύρια προστίθενται σε αυτά από μεταφορά μέσα στο τμήμα 3. Αυτά θα δοθούν για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, ιδιαίτερα για τα άμεσα μέτρα αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών. Νομίζω αυτά θέλατε να μάθετε. Ναι, σας ευχαριστώ. Για το 13 ή το 14. 13. Το 13 ως προβλέψεις. Ως προβλέψεις. 13. για το ερώτημα Λαβία για τον διορθωτικό προπολογισμό 8 και την προσαρμογή των 14,7 δις από το Συμβούλιο. Αυτό είναι η άποψη του Συμβουλίου και θεωρεί ότι πρόκειται για μια προσαρμογή που ανταποκρίνεται στη διαφωνία που υπάρχει για τη συμπερίληψη στον προϋπολογισμό, για τον συνυπολογισμό των πληρωμών και τον τρόπο κατανομής του Ταμείου Αλληλεγγύης. Πρέπει να το δούμε και αυτό. Εν καιρό το δέοντι. Υπάρχει όμως μια δυσκολία που σχετίζεται με τον διορθωτικό εννέα. Τώρα, για αυτόν θα ήθελα να πω στην κυρία Ολμέγερ ότι και εγώ θα ήθελα να βρω 200 εκατομμύρια για τις σφαιρικές μεταφορές λέω ε. και εγώ θα ήθελα να βρω 200 εκατομμύρια για να υπάρχουν περισσότερα χρήματα στις πληρωμές για την έρευνα. Ήταν μεγάλη τύχη σε εισαγωγικά όταν προετοιμάζαμε αυτή τη σφαιρική μεταφορά ότι υπήρχαν 289 εκατομμύρια από στο πρόγραμμα. Αν δεν είχαν υπάρξει αυτά τα 289 εκατομμύρια που μας εξέπληξαν όλους πολύ ευχάριστα, τότε η σφαιρική μεταφορά θα ήταν μόνο 220 εκατομμυρίων, δηλαδή η χαμηλότερη ιστορικά που έχει ποτέ σημειωθεί στην ιστορία του προϋπολογισμού της Ένωσης. 200 εκατομμύρια λοιπόν, πού να βρεθούν, ψάχνουμε κι εμείς, Κάνουμε ό,τι μπορούμε, είμαστε διατεθειμένοι να τα βρούμε και ψάχνουμε μήπως υπάρχουν και πουθενά αλλού κρυμμένοι τέτοιοι θησαυροί. Αμφιβάλλουμε όμως, γιατί ήδη με μεγάλη δυσκολία καταφέραμε να πετύχουμε αυτή τη σφαιρική μεταφορά τώρα για τον διορθωτικό εννέα. Είναι σαφές ότι Αν τα 409 εκατομμύρια χρησιμοποιηθούν για χρηματοδότηση του, τότε μένουν μόνο άλλα 100 από την σφαιρική μεταφορά, για τη σφαιρική μεταφορά. Και είναι απολύτως απαραίτητο να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε όλα τα κονδύλια που χρειάζονται για τους πρόσφυγες Συρία, από τη Συρία. Ξέρετε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα πληρωμών για τα επίγοντα μέτρα βοήθειας, την ανθρωπιστική βοήθεια για τους σύρους πρόσφυγες, μόνο 70 εκατομμύρια και γι' αυτό, αυτό σημαίνει ότι 31 εκατομμύρια σύνολο έχουν μείνει για τη χρηματοδότηση. Δηλαδή λίγα. Και η Κομισιόν θεωρεί ότι υπό τη Άφταση συνθήκας θα έπρεπε να δώσουμε προτεραιότητα στις πληρωμές που ωφελούν εκείνους που αν δεν τους πληρώσουμε θα χρειαστεί να τους αποζημιώσουμε ή να πληρώσουμε πρόστιμα για καθυστέρηση. Θα τους δώσουμε λοιπόν αυτούς προτεραιότητα στην κινητοποίηση των κονδυλίων. Τώρα, τι γίνεται με το ότι η ψηφοφορία για τους διορθωτικούς 6 και 7 δεν θα μπορέσει να γίνει παρά στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Η Ολομέλεια εκείνη αρχίζει 19 Νοεμβρίου και ο κανονισμός για τη διάθεση των ιδίων πόρων είναι σαφής. Λέει δηλαδή ότι εάν εγκριθεί ο προϋπολογισμός μετά τις 15 του μήνα, τα χρήματα θα διατεθούν στην Κομισιόν την πρώτη εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα, του μήνα μετά την ψηφοφορία του μήνα νήσιν ένα δηλαδή. αν η ψηφοφορία γινόταν πριν τις 15 Νοεμβρίου θα δινόταν τα χρήματα την 1η Δεκεμβρίου. Ενώ στις 19 Νοεμβρίου 2 Ιανουαρίου θα διατεθούν τα χρήματα. Αποτέλεσμα η Κομισιόν θα έχει πολύ σοβαρά προβλήματα για τις πληρωμές. Υπάρχουν τα κονδύλια, αλλά δεν έχουμε το ρευστό για να τα πληρώσουμε. Και άρα το πιο πιθανό είναι, σίγουρο μάλλον, είναι ότι θα υποχρεωθούμε να αναστείλουμε τις πληρωμές αυτές ή να τις αναβάλουμε για αργά το Νοέμβριο αυτό να αναστείλουμε τις πληρωμές. Αυτά είναι, αυτή είναι η κατάσταση, έτσι παρουσιάζεται. Μας ανησυχεί πολύ σοβαρά για τις επιπτώσεις που θα έχει. στους ανθρώπους αυτούς που έπρεπε κανονικά να ωφεληθούν. Αλλά σας τα λέω ειλικρινά για να ξέρετε πώς ακριβώς έχουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γενικέ Διευθυντά. Από ό,τι κατάλαβα λοιπόν για το ερώτημα που είχα θέσει, 30 περίπου εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για, τα, για τη Λαμπεντούζα μετά από μεταφορές που αφορούν προβλέψεις του 13 και οι πληρωμές θα γίνουν στο τέλος του χρόνου και θα συμπεριληφθούν δεν θα μπουν στον προϋπολογισμό του 2013. Αυτό ήθελα να ξέρω. Λοιπόν, επίσης κατάλαβα, χωρίς να με κλείσει αυτό βέβαια, αλλά είναι καλό που το είπατε δημόσια, ότι εάν παραμείνουμε στη θέση του Συμβουλίου όπου να χρηματοδοτηθεί ο διορθωτικός 9 εξ ολοκλήρου με την σφαιρική μεταφορά, με τα 400 εκατομμύρια δηλαδή, αν παραμείνουμε σε αυτό, τότε για να μιλήσουμε ομά αλλά ρεαλιστικά, θα χρειαστεί να επιλέξουμε μεταξύ ή να θυσιάσουμε τους σύρους πρόσφυγες ή να μην εφαρμόσουμε τον προϋπολογισμό. Γιατί αν υποχρεωθούμε να πληρώσουμε για τις καθυστερήσεις αυτό θα σημαίνει ότι η Κομισιόν δεν έχει εφαρμόσει τις διορίες που προβλέπονται κανονικά από το δημοσιονομικό κανονισμό. Θα τα δουν αυτά και οι εισηγητές βέβαια γραμμή γραμμή, αλλά να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι παίζεται. Πρέπει κάποτε κάποια στιγμή το κάθε όργανο να αναλάβει τις ευθύνες του. Για δε τις καθυστερήσεις στη λήψη των αποφάσεων, υπενθυμίζω ότι η καθυστέρηση αυτή, χωρίς να επιμένω, δεν αρχίζω το blame game εδώ πέρα, γιατί δεν είχε νόημα, υπενθυμίζω απλώς ότι ο διορθωτικός προϋπολογισμός 6 2,7 δισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια πρόσθετων πόρων από την εισφορά κτλ. που πληρώνουν επομένως τα κράτη-μέλη και που είναι τελείως απαραίτητος λόγω της ύφεσης και της μείωσης από τα έσοδα από τα τελωνία. δεν έχει ακόμη εγκριθεί από το Συμβούλιο. Ούτε μας έχει υποβληθεί εμάς. Και το Συμβούλιο δεν θέλει να τον εγκρίνει εν καιρός. Επομένως υπάρχει ένα πρόβλημα αρεστότητας το οποίο φταίει 100% το Συμβούλιο. Για σοβαρούς λόγους. Για σοβαρούς λόγους δεν λέω. Αλλά πάντως το Συμβούλιο καθόλου δεν το έθιξε αυτό το θέμα. Καθόλου. Επίσης, δεν θα είχε καθόλου κανένα αποτέλεσμα να προχωρήσουμε με τον διορθωτικό προϋπολογισμό υπαριθμών 8 με το Συμβούλιο, διότι ούτως ή άλλως δεν θα είχαμε μπορέσει να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια επί του διορθωτικού προϋπολογισμού 8 και δεν θα είχε τα 3,9 δις ε, η Κομισιόν γιατί το Συμβούλιο έτσι που τα κατάφερε και δεν το καταλαβαίνω αυτό καθόλου το Συμβούλιο λοιπόν τα κατάφερε να μην μπορέσει να ψηφίσει στο χρονοδιάγραμμά του για το διορθωτικό προϋπολογισμό υπαριθμών 8 πριν την 30 Οκτωβρίου. Ακατανόητο. Επομένω, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, το Συμβούλιο αποφασίζει. Είμαστε στα χέρια του Συμβουλίου. Για την ώρα δεν κατηγορούμε κανέναν για τίποτε. Αλλά, αλλά εάν ε, κάποιοι παραπονεθούν, θα πρέπει τα παράπονά τους στο Συμβούλιο να τα κάνουν. Λαμβάνοντα υπόψη τα όσα ελέγχθησαν. Καλό τους ε, εισηγητέ, ε, το κάνουν ήδη, αλλά εν πάση περιπτώσει του ενθαρρύνω περαιτέρω, να ε, δουν τα πράγματα με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, να δουν ποιες είναι οι γραμμές οι οποίες επηρεάζονται από, το, τη συνολική καταβολή, να δουν γραμμή προς γραμμή ε, ε, ποια είναι η θέση του Συμβουλίου. Ξέρουμε ότι το Συμβούλιο όσον αφορά να, ε, όσον αφορά τη συνολική καταβολή θέλουν, ε, θέλει το Συμβούλιο λέω, να δώσει τα 400 εκατομμύρια στο διορθωτικό προϋπολογισμό. Τι θα γίνει με τα 109 εκατομμύρια, αυτά τα 100, τα 100 ε, από τα, υπόλοιπα μάλλον συγγνώμη όπως έλεγε και η Μόνικα να δώσουμε 100 εκατομμύρια για την έρευνα γίνεται αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένη όσον αφορά αυτή την συλλογική διαπραγμάτευση. Ο Ναράγχο, παρακαλώ Ναράγχο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, το Πρόεδρο και όσους εργάστηκαν ε, σκληρά σε αυτό το θέμα και μας έδωσαν εκτενή αναφορά. Εγώ θα μιλήσω πολιτικά ε, γιατί είμαστε σε πολιτικό χώρο. Μας ανακοινώσατε, αν, κατάλαβα καλά, ότι αποφάσισε η διάσκεψη των Προέδρων να αναβληθεί η απόφαση για τον Νοέμβριο για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Σωστά το κατάλαβα. Ωραία. Και αυτό τι είναι τώρα, είναι οριστικό, μετάκλητο, αλλάζει, ανατρέπεται, τι γίνεται. Επίσημα μπορούμε να προχωρήσουμε, γιατί βλέπω δύο ε, ειδών προβλήματα ένα πολιτικό και λυπάμαι πάρα πολύ για αυτή την απόφαση, γιατί εμείς τι μήνυμα στέλνουμε στους συμπολίτε μας, ότι για άλλη μια φορά ερχόμαστε να ρίξουμε περισσότερο μύχλη και καπνό σε ένα πρόγραμμα και ένα πρόβλημα που έπρεπε να έχει λυθεί ή την άλλη εβδομάδα και από την άλλη υπάρχει και ένα πρόβλημα δημοσιονομικό πέρα από το πολιτικό που συνδέεται με όλους τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς που πολύ ωραία μας εξήγησε ο Τζοβάνι Λαβία. Γιατί κάθε διορθωτικός έχει ε, το δικό του δρόμο προς την επίλυση. Βία στα ισπανικά που είναι και λογοπαίγνιο με το λαβία. Η διάσκεψη των Προέδρων μπορεί να έδωσε νομικά επιχειρήματα και δημοσιονομικά αλλά είναι αρκετά γερά. Από πλευράς δημοσιονομικής μπορεί να λύνονται τα προβλήματα, αλλά και από πλευράς νομικής επίσης. Γιατί είχαμε λίγο σκοντάψει σε σημαντικά θέματα και σημαντικούς κανονισμούς, όπως είπατε και εσείς, Πρόεδρε, αλλά πολιτικά πρέπει να πω ότι θλίβομαι από την απόφαση αυτή. Και υπήρχε δυνατότητα επίληψης σε αυτό το χρονικό ορίζοντα. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα να εξηγήσει στους πολίτες ότι σηκώνει τα χέρια ψηλά, ότι δεν μπορείς να λύσεις τέτοια προβλήματα που είναι διαδικαστικά. Το ξέρω ότι υπάρχει και δικονομία στο δίκαιο ε, και το χρησιμοποιούν ορισμένοι και για να χρονοτριβούν και για να παρακολύουν τις διαδικασίες επί της ουσίας, αυτά τα δικολαβίστικα, αλλά επί της ουσίας νομίζω ότι είναι κάπως δύσκολο να βγω να αντιμετωπίσω τους πολίτες και να πω ότι ξέρετε είναι πάρα πολύ περίπλοκα τα πράγματα, οι διαδικασίες. Ε, όχι ουσίας, επαναλαμβάνω διαδικασίας και χρονοτριβούμε, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε για να δώσουμε το ok. Ε, εκεί που βρισκόμαστε πρόεδρε, αυτό που χρειαζόμαστε είναι σταθερότητα και ένα μήνυμα ηρεμίας, ησυχίας χρειάζονται οι πολίτες και οι θεσμοί που είναι τελικά δικαιούχοι ε, της ε, κοινοτικής χρηματοδότησης. Εμείς θέλουμε το αντίθετο μήνυμα. Τους έχουμε μπερδέψει τους ανθρώπους ε, όλο αυτό το γαπνό και την ομίχλη που ρίχνουμε στα πράγματα. Το ξέρω ότι είναι πολιτική απόφαση και μας εξήγησε ο Γενικός Διευθυντής τα προβλήματα που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τα βγάλει πέρα στον προϋπολογισμό και ε, στη συνολική μεταφορά πιστώσεων. Εγώ σας μιλώ πολιτικά, γιατί αυτό είναι απόκειται στην Επιτροπή μας που είναι πολιτικό όργανο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητές συνάδελφοι. Στη διάσκεψη των Προέδρων είπα ότι από πλευράς Επιτροπής Προϋπολογισμών ε, θεωρούμε ότι είναι χρήσιμη ακόμα η ημερομηνία της 23ης Οκτωβρίου. Όμως δεν αποφάσισε κατά αυτήν την έννοια η διάσκεψη των Προέδρων. Και δεν θα αλλάξει αυτή η απόφαση. Όμως αγαπητέ μου φίλε, το πρόβλημα δεν είναι διαδικαστικό εδώ και δεν, ε, ε, το, το λάθος ε, δεν αφορά το Κοινοβούλιο. Πώς θέλετε να ψηφίσει το Κοινοβούλιο επί ενός κειμένου επί του οποίου δεν έχει ψηφίσει το Συμβούλιο ακόμα. Ναι, βεβαίω υπάρχει καθυστέρηση, αλλά δεν ευθύνεται για αυτήν το Κοινοβούλιο. Και γιατί δεν ψήφισε το Συμβούλιο, παρακαλώ, γιατί κάποιε χώρε μέλη δεν θέλουν ή δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Ιδού και δυστυχώς δεν μπορούν να ψηφίσουν λοιπόν το δικό σας προϋπολογισμό και το δικό μας προϋπολογισμό. Εάν θέλουμε να μιλήσουμε με πολιτικούς όρους, αυτή είναι η κατάσταση, αλλά το σύστημα είναι τέτοιο που επιτρέπει σε κυβερνήσεις σε κάποιες κυβερνήσεις να κρυφτούν πίσω από αυτή την απόφαση. Τα θέματα τα οποία μας απασχολούν εδώ ε, ε, προσμετρώνται σε δισευρώ, Αφορούν ε, ε, την κοινωνική πολιτική, την ανθρωπιστική βοήθεια, ε, την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, πράγματα ζωτικής σημασίας. Αλλά από πλευρά Συμβουλίου τελικά προκαλούν μονάχα συζητήσεις και κλεισμένων των θυρών σε επίπεδο υψηλόβαθμων υπαλλήλων. Δεν ξέρουμε τι γίνεται πίσω από αυτές τις κλειστές πόρτες. Ε, και μετά στα συμβούλια αυτά είναι σημεία α. Και επομένως ε, και κλεισμένο των θυρών, χωρίς δημοσιογράφους, χωρίς κάμερες και όταν μετά σκοντάψει η διαδικασία λένε «Α, φταίει το κοινοβούλιο». Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η, κυβέρνηση δεν είναι στη χώρα μου, δεν είναι του, δικού μου πολιτικού σχηματισμού, αλλά και όταν είμαστε εμεί, α πούμε, στην κυβέρνηση, το ίδιο έκανα. Καταδίκαζα, κατήγγελα τι αποφάσει αυτέ και τι διαδικασίε αυτέ. Αύριο θα πρέπει να αποφασιστεί ε, πότε οι κυβερνήσεις των χωρών μελών επιτέλους θα αναλάβουν τις ευθύνες τους, θα κάνουν ε, τις ψηφοφορίες που πρέπει να κάνουν. Γιατί οι διαδικασίες είναι συγκεκριμένες. Πρώτα γίνεται η ψηφοφορία στο Συμβούλιο και μετά γίνεται η ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο. Προσθέτω δε ότι Εάν δεν είχε τροποποιηθεί η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όλα τα προβλήματα πληρωμών του 2013 θα είχαν ε, διευθετηθεί από τον Ιούνιο του 2013. Γιατί το Κοινοβούλιο στις διαπραγματεύσεις του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου είχε πει δέχομαι τα αριθμητικά στοιχεία έστω και αν είναι πολύ χαμηλότερα από ό,τι ήθελα και έστω και αν έχουν μειωθεί περαιτέρω. Δέχομαι λοιπόν τους αριθμούς, αλλά ε, επιβάλλω κάποιες προϋποθέσεις. Να εκτελεστεί ο προϋπολογισμός του 2013 σύμφωνα με τις συνθήκες, ε, με όλες τις υποχρεώσεις που είχαν αληφθεί, με πληρωμή όλων των ε, καταβολών που είχαν αποφασιστεί για το 2013 έτσι ώστε η κατάσταση να είναι υγιής. Η Κομισιόν ήδη τότε ε, έκανε μια εκτίμηση της τάξης των 11,2 δις που θα έπρεπε να προσθεθούν στο 2013 και το Κοινοβούλιο στήριζε τη θέση αυτή και ζητούσε λοιπόν 11,2 δις. Εκείνη την εποχή το Συμβούλιο λόγω των δυσκολιών που αντιμετώπιζαν κάποιες ε, κυβερνήσεις τις οποίες γνωρίζουμε κι εσείς κι εμείς δέχτηκε μία πρώτη τρανς 7,3 δις και μας είχε υποσχεθεί τα υπόλοιπα. Α, το Συμβούλιο λέει ίσως θα έχετε και τα 3,9 αλλά παρόλα αυτά από εκεί θα σας αφαιρέσω 400 εκατομμύρια. Αυτή είναι η κατάσταση. Πολιτική συμφωνία η οποία αμφισβητείται. Εγώ την υπογραφή που βάζω σε, σε, στις ε, συμφωνίες και στις συμβάσεις ε, την τιμώ την υπογραφή μου ενώ το Συμβούλιο δεν είναι το ίδιο. Βάζει την υπογραφή του και μετά αλλάζει τις προϋποθέσεις. Γιατί, ε, αλλά πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό γιατί διαφορετικά το Κοινοβούλιο δεν αξίζει τίποτα και τελικά βάζει απλώς τη βούλα στις αποφάσεις του Συμβουλίου. Και μετά όταν ε, δεν, αρέσει, δεν αρέσουν οι αποφάσεις τότε όλοι οι σκανδαλισμένοι λένε μα το Κοινοβούλιο τι έκανε, το Κοινοβούλιο φταίει κτλ. Δεν είναι έτσι όμως. Θα πρέπει να πάρουμε θέση όσον αφορά τα θέματα αυτά. Και για να πάρουμε θέση θα πρέπει να έχει ψηφίσει το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο λοιπόν αργή καθυστερεί 2,7 ε, ε, ε, δις ευρώ που αφορούν τον διορθωτικό προϋπολογισμό 6 και που αντλούνται από τους ίδιους πόρους για τον απλούστατο λόγο ότι ορισμένες χώρες αντιμετωπίζουν δυσκολία να ε, ε, δώσουν ε, τις συνεισφορές τους και θα μετακυλιστεί ας πούμε ε, η εισφορά τους από το 2013 στο 2014 και το Συμβούλιο, δηλαδή οι κυβερνήσεις δεν έχουν το θάρρος και την τόλμη να το εξηγήσουν αυτό στην κοινή γνώμη. Εμείς κατανοούμε ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν μεγάλη δυσκολία τούτη τη στιγμή να αυξήσουν τη συνεισφορά τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα έπρεπε να έχουν το θάρρος να το συζητήσουν, να το καταθέσουν αυτό στη δημόσια συζήτηση. Εν τω μεταξύ βεβαίως καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να δεχτεί οποιαδήποτε κατηγορία και βεβαίως δεν πρέπει να έχει καμία ενοχική στάση για τα όσα συμβαίνουν. Έχουμε εδώ δαπάνες οι οποίες δεν θα μπορέσουν να καταβληθούν έγκαιρα σε πολύ κακή στιγμή και σε, σε, σε τομείς οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι ανθρωπιστικοί τομέα, κοινωνική πολιτική κτλ. Κύριος Χάρτονγκ, Πρόεδρε, ο αξιότιμος συνάδελφος του ΕΛΚ μόλις είπε ότι δεν μπορούμε πια να τα εξηγήσουμε στους πολίτες μας. Και συμφωνώ απολύτως. Τι να ε, εξηγήσουμε σε αυτά τα ντάπ και τα δισεκατομμύρια που κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά. Χάος, σκέτο. Το είπατε κι εσείς η πολιτική λύση κανονικά θα ήταν απλή. Να κλείσουμε τα αερολά, να κατεβάσουμε, να βάλουμε λουκέτο και να δώσουμε στα κράτη-μέλη ξανά αυτές τις αρμοδιότητες. Πολλά λεφτά χάνουμε με αυτή την πολιτική. Πρόεδρε, θέλω να τονίσω ε, ότι ε, ε, πολιτικά αυτά τα πράγματα εγώ δεν μπορώ να τα ακολουθήσω. Δεν ανθέβαλα έτσι σας ε, διαβεβαιώ. Λοιπόν, δύο κόμμα έχουν ζητήσει το λόγο και μετά να ψηφίσουμε. Γιατί λέει εδώ ώρα ψηφοφορία. Ε, Γιούτα Χάουκ. Ο Αλέν τα εξήγησε εκτενέστατα και πολύ καλά και μπορούμε να βγούμε προς τα έξω και να τα εξηγήσουμε σε κάθε πολίτη. Γιατί είναι σχετικά σαφή όλα αυτά και απλά. Αυτό που είπατε ότι τα τάπ είναι ένα χάος διοικητικό είναι λάθος. Δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτό ε, το λάθος μονοπάτι. Οι διορθωτικοί προϋπολογισμοί είναι το αποτέλεσμα αυτού που μας κάνει το Συμβούλιο εδώ και δύο χρόνια. Κάθε φορά μας αναγκάζει ε, οι πληρωμές να είναι πολύ λίγες, πολύ λίγες πληρωμές. Τα δύο τελευταία χρόνια θα μπορούσαμε ήδη πριν από δύο χρόνια και θα έπρεπε να το είχαμε κάνει, να αρνηθούμε, δεν το κάναμε γιατί έχουμε πολιτική υπευθυνότητα και γιατί χρειαζόμαστε προπολογισμό και η Κομισιόν τα ίδια λέει. Και είδαμε που οδηγηθήκαμε τώρα ότι χρειαζόμαστε ένα σωρό DAPs, πραγματικά διορθωτικούς προϋπολογισμούς και να ξαναβάζουν πάντα το χέρι στην τσέπη τα κράτη-μέλη. Και αυτό που λέει ολα ειναι είναι σωστό. Ορισμένα κράτη-μέλη έχουν δυσκολίες, τι να κάνουμε. Και μπορούμε να το κατανοήσουμε αυτό και πιστεύω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ορισμένα κράτη-μέλη μπορεί να βρει ε, κάποιες τεχνικές λύσεις τα χρήματα που πρέπει να καταβληθούν να δοθούν σε δόσεις λίγο αργότερα, τρόπος υπάρχει. Πάντως είναι σαφές επίσης ότι τουλάχιστον μια χώρα κράτος μέλος που είναι υπεύθυνη για ένα πέμπτο του κοινοτικού προϋπολογισμού δεν έχει δυσκολίες και μπορεί να τα δώσει και πρέπει να τα δώσει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχει δυσκολίες. Και αυτή είναι ακριβώς εκείνη ε, που, γιατί ακούμε και φήμες από το Συμβούλιο, είναι εκείνοι που χρονοτριβούν και τώρα ζήτησαν τον ΤΑΠ 8 να συνδεθεί με το 9 προφανέστατα και μόνο εάν ε, το DAP9 ε, πληρωθεί από τη μεταφορά των πόρων θα συμφωνήσουμε. Και ποιοι είναι αυτοί οι Γερμανοί, να το πω έτσι. Οι Γερμανοί το ξεκίνησαν αυτό. Και όλοι οι υπόλοιποι, τα υπόλοιπα 4 πέμπτα του προπολογισμού, που είναι 27 ε, δόσεις, 27 φέτες, άφησαν τη Γερμανία να τους εκβιάσει. Και είπανε αφού του λέει Γερμανία, Μα τι ανοησίες είναι αυτές. Και μετά βγαίνει ο Γερμανός πρέσβης και λέει και η Προεδρία του Συμβουλίου ότι θα πρέπει να τα διαβιβάσει στον Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών διεπιστολής, με αλληλογραφία και μετά τελειώνει η υπόθεση. Μα τι ε, αντίληψη έχουμε για τη δημοκρατία να πάρει ευκή. Εμείς δεν φταίμε ε, που είναι χάος, αν είναι χάος ο προϋπολογισμός. Και πραγματικά, μην με παρεξηγείς, ξέρω ότι είσαι σε δύσκολη θέση γιατί το κόμμα σου κυβερνάει στην Ισπανία, λέω αυτά στον Αράχο. Ε, εμείς είμαστε στο απέναντι στις κυβερνήσεις, είτε αυτές είναι τώρα συντηρητικές, φιλελεύθερες ή σοσιαλιστικές. Αυτά. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να αποφύγουμε μάλλον να κάνουμε εδώ θεωρήσεις έτσι πολιτικής πολιτική. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ναράχο. Μα δεν είχα εγώ καμία τέτοια πρόθεση. Ένα μήνυμα ήθελα να σας πω. Έχουμε βρεθεί σε μια κατάσταση. Το κοινοβούλιο το οποίο είχε συνεπή και έξυπνη στάση μέχρι εδώ ε, χρεώνεται διάφορα πράγματα. Εγώ δεν ήθελα να το προσάψω στο κοινοβούλιο αυτό σε καμία περίπτωση. Απλώς να διαβιβάσω στους συναδέλφους ότι αυτές οι ανεπιθύμητες συνέπειες και οι παρενέργειε ε, της διαδικασία αυτής που διονύζεται είναι πάρα πολύ αρνητικέ για τον κόσμο. Εγώ δεν ακολουθώ εντολέ τη κυβέρνηση μου, τουλάχιστον προσωπικά, ακριβώς πιέζω προς την κατεύθυνση που λέτε και που εξηγήθηκε εδώ. Δηλαδή ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του και να καταβληθούν οι πληρωμές από όλες τις κυβερνήσεις για να τελειώνει το πρόβλημα και να λυθεί. Δεν ξέρω αν σας έδωσα την εντύπωση αυτή, δεν ήταν καθόλου πρόθεσή μου να βγάλω κανένα λόγο εδώ ότι α, όχι, σε καμία περίπτωση. Τίποτα δεν είναι πιο μακριά από αυτές τις προθέσεις. Δεν θεωρώ ότι το αρπηλίζει το κοινοβούλιο την κατάσταση. Το αντίθετο. Ήθελα να πω αν υπάρχει δυνατότητα να απεγκλωβιστεί αυτή η ιστορία και να δοθεί μια θετική κατεύθυνση από δική μα πλευρά να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εδώ στο δημοσιονομικό πλαίσιο έχουμε πετύχει πολλά. Μεταξύ αυτών και ο μηχανισμός που πραγματικά είναι σημαντικός. Και ποιος είναι αυτός απλούστατα το γεγονός ότι ανοίγει η πόρτα για να μπορέσουν στους ιδίους πόρους ε, στο μέλλον να υπάρξουν εξελίξεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και σημαντικότατος πυλώνας και το κάναμε εμείς, το καταφέραμε εμείς. Μπορούμε το ε, πολιετές να το εγκρίνουμε. Και οποιαδήποτε καθυστέρηση είναι δύσκολο να την εξηγήσουμε στην κοινή γνώμη. Εγώ καθόλου όμως δεν ήθελα να σας δώσω την εντύπωση ότι φταίει το κοινοβούλιο. Και είναι ένα στοιχείο που βοηθάει στην κολυσιεργία. Το αντίθετο. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους σας για τη δουλειά που κάνατε όλο αυτό το χρόνο και εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πρόσληψη λίγο να απαντήσω στην αγαπητή μου συνάδελφο και φίλη Γιώτα γιατί επευθύνθηκε σε μένα προσωπικά. Ευχαριστώ πολύ. No, Σας ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνουμε, καταλαβαίνουμε και άλλωστε νομίζω ότι θα πρέπει να αποφύγουμε να κατηγορήσουμε τη μία ή την άλλη χώρα. Δεν ωφελεί αυτό τίποτα. Ξέρουμε ποιοι είναι οι συνήθεις ύποπτοι. Υπάρχει και ένας που είναι πιο συνήθις από τους άλλους. Μεταξύ των υπόπτων ε, και μετά έχουμε και όλους τους συνήθεις υπόπτους που είναι οι ε, καθαροί συνεισφορείς. Ξέρουμε, ξέρουμε ποιες είναι οι συσχετισμοί δυνάμεων, ποιοι είναι οι συσχετισμοί δυνάμεων στο Συμβούλιο των Υπουργών. Όταν υπάρχει μια χώρα η οποία ζητάει κάτι παραπάνω από τις άλλες ε, και επιμένει περισσότερο, ξέρουμε ότι πίσω του κρύβονται άλλες χώρες ή και άλλες χώρες δεν είναι δικός μας ρόλος του Κοινοβουλίου να κατηγορήσει τη μία ή την άλλη χώρα, αλλά εμείς σαν Κοινοβούλιο οφείλουμε να υπεραμηθούμε των ε, συμφερόντων ε, και των ε, πολιτών και που βέβαια και στόχος μας είναι και, και ρόλος μας είναι να ελέγχουμε την κατάσταση όσον αφορά τις ε, κυβερνήσεις ας πούμε και ε, το τι κάνει το Συμβούλιο. Από την άλλη πλευρά όμως επιμένω ότι δεν είναι δυνατόν να κατηγορούμαστε εμείς για τις ε, καθυστερήσεις και τις όποιες επιπτώσεις η Άλτα. Τελευταία ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μέχρι τώρα Έχουμε συζητήσει και έχουμε πληροφορήσει όλα τα μέλη της Επιτροπής μας για τα τελευταία τεκτενόμενα. Είναι σημαντικό να ξέρουμε τι έγινε στην διαπραγμάτευση για να ξέρουμε και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις, όχι μονάχα οι πολιτικές επιπτώσεις αλλά και οι πρακτικές άμεσες επιπτώσεις και πώς αυτές οι επιπτώσεις θα διαμορφώσουν ε, την, ε, την, ε, το χρονοδιάγραμμα και το θεματολόγιο των επομένων, του επομένου διαστήματος το Κοινοβούλιο, συμφωνώ και εγώ, ότι δεν πρέπει να ε, υποχωρήσει ε, σε, αυτή, σε αυτόν τον εκβιασμό ε, του Συμβουλίου που θα μπορούσε να μας πιέσει για να κάνουμε άσχημα τη δουλειά μας. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε το σκεπτικό λίγο παραπέρα. Το ζήτημα είναι πολιτικό και αφορά ε, και τις επιλογές ε, του Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο λέω εξ αρχής ότι δεν πρέπει να υποχωρήσει στους εκβιασμούς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με όλες τις επιλογές του Κοινοβουλίου. Η ομάδα μου δεν συμφωνεί ε, κυρίως με την συμφωνία που έκανε το Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Γνωρίζετε ότι η πολιτική μου ομάδα δεν συμφωνεί με αυτήν την πολιτική συμφωνία για πολλούς λόγους διότι το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι ένα πλαίσιο το οποίο δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις στις οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη, ε, κυρίως δε σε χώρες που όπως η δική μου ε, βρίσκονται ε, κάτω από την επιρροή της Τρόικα και που ε, ε, ε, αναγκάζονται, τους επιβάλλονται μέτρα, αναγκάζονται να λάβουν μέτρα τα οποία όχι μόνο δεν προωθούν την ανάπτυξη αλλά οδηγούν και σε αντικυκλικές επιπτώσεις που επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο και τις κοινωνικές δυσκολίες και την ανεργία των νέων κτλ. Οι πολιτικές λιτότητας ε, οι οποίες εφαρμόστηκαν ε, από τις ε, διάφορες κυβερνήσεις μετά από εξαναγκασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οδήγησαν στα όποια προβλήματα και τώρα περάσαμε από την υποχρεωτική λιτότητα στην, στον εκβιασμό. Ε, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι διατρέχουμε σοβαρό κίνδυνο τελικά να βγούμε από αυτή την κατάσταση όλοι εξαιρετικά αποδυναμωμένοι και οι κυβερνήσεις ε, και οι πολίτες και τα λοιπά. Δηλαδή ε, και αποδυνάμωση όλων λόγω αυτού του εκβιασμού απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και μεγάλες απώλειες σε κάθε επίπεδο για τους πολίτες. Θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω ουσιώδεις, βασικές αμφιβολίες οι οποίες δεν συνδέονται ε, με την ίδια τη διαπραγμάτευση, με τον ίδιο τον ε, προϋπολογισμό. Ε, η ένστασή μας είναι ότι οδηγούμεθα σε μια Ευρώπη de σε μια Ευρώπη η οποία θα αρκείται στα ελάχιστα. Αυτό καταλαβαίνετε ότι μας πάει πάρα πολύ πίσω οι πιο ασθενείς δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν εν τέλει. Αυτή η Ευρώπη που κλείνεται όλο και περισσότερο απέναντι σε αυτούς που προσπαθούν να περάσουν τα σύνορά της. Ε, είναι μια Ευρώπη η οποία κλείνεται ακόμα και απέναντι στους δικούς της τους πολίτες. Αναφέρομαι στα όσα περνάει η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή αναφέρομαι σε τραγωδίες τύπου Λαμπεντούζα. Είναι καταστάσεις οι οποίες αντικατοπτρίζουν ε, αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι εδώ η ε, ε, ευθύνη του Κοινοβουλίου είναι μεγάλη. Οι μεγάλες ε, ομάδες δέχτηκαν το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και αυτό οδήγησε σε αδιέξοδα και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιστρέψουμε στην αρχική κατάσταση με αυτό το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Εκφράσατε σαφώς την άποψη της πολιτικής σας ομάδας και πρέπει να πω ότι πολλοί μεταξύ ημών συμφωνούμε με πολλά από τα σημεία αυτής της διάγνωσης που κάνατε. Τώρα, για... πρέπει να αρχίσουμε την ψηφοφορία. Ευτυχώς, αλλά έχουμε τις μισές ψηφοφορίες που ακυρώθηκαν και προτείνω να αρχίσουμε από το 20. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Έτηση από την Κομμουνιδάδ Βαλενθιάνα. Εισηγητής είναι ο συνάδελφός μας ο Πλένκοβιτς. Έχετε τους καταλόγους ψηφοφορίας, εγώ δεν τον έχω λέει ο πρόεδρος, αλλά θα βρω. Θα το βρω. Έκθεση λοιπόν Πλένκοβιτς με ορισμένες τροπολογίες. Έχετε όλες τις κάρτες σας. Ο κύριος Πλένκοβιτς δεν θα ψηφίσει ο ίδιος. Όχι θα ψηφίσει, θα ψηφίσει. Λοιπόν, υπάρχουν οι πατροπολογίε των ίδιων πάντοτε συντακτών Μπερές και άλλων δηλαδή επί των οποίων συμφωνεί ο εισηγητής. Είναι τροπολογίες 1, 2, 3, 4, 6 γιατί η πέμπτη καλύπτεται ήδη. Όλες μαζί, όχι, ναι, όχι. Γιατί αν θέλετε να αφαιρέσετε μία από αυτές τις τροπολογίες. Ένα και δύο. Μαζί της ένα και δύο δηλαδή. Ένα και δύο. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Τέσσερις. Αποχές εγκρίνονται. Μαζί επίσης τρία, τέσσερα και έξι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Των φιλελευθέρων οι 7, ο ψυχητής είναι κατά υπέρ, 3 κατά. Οι μεγάλες ομάδες και οι φιλελεύθεροι αποχές, ο κύριος Αρτών. Απορρίπτεται. 8. Ο συγητής είναι κατά, υπέρ. Η ομάδα του συγητή. Α, όχι. Λοιπόν, κατά οι υπόλοιποι αποχές απορρίπτεται. Τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ηλεκτρονική. Α, δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει το μηχάνημα. Président, voilà.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 Ξανά, τώρα δουλεύει. Δεν έχει ψηφίσει κάποιος. Α, 21, εντάξει. 20 υπέρ, 1 κατά. Καμία αποχή, συγχαρητήρια. Τώρα, τώρα έκθεση Χάουγκ. σιδηρόδρομοι. Δύο τροπολογίες της εισηγήτριας, η τρία και τέσσερα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία πέντε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται για το ψήφισμα. Δύο τροπολογίες της εισηγήτριας ένα και δύο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Ηλεκτρονική και τελική ψηφοφορία. Να δούμε αν δουλεύει στο μηχάνημα. Δουλεύει. Ψηφίστε. Ωραία ψήφισαν όλοι. Έληξε. 20 υπέρ. Μία ψήφος κατά. Εγκρίνεται. Η άλλη έκθεση. Η άλλη Ορίστε Γιούτα. Κοιτάξτε, ξέρω ότι δεν συνηθίζεται, αλλά επειδή συζητήσαμε και ακούσαμε τις αντιρρήσεις της Επιτροπής Ήτρε, προτείνω κύριε Πρόεδρε, για προφορική τροποποίηση να προτείνουμε κάτι για την παράγραφο 6 να μείνει ως έχει αλλά στο τελευταίο της μέρος να προσθέσουμε τη συζή ή να τροποποιηθεί το μπερέκ ανάλογα με κτλ. Ξέρω κύριε Πρόεδρε ότι δεν συνηθίζονται τέτοια πράγματα. Αλλά να. Δεν λέω ότι πρέπει τελείως να τα κλείσουμε όλα, αλλά ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε εδώ μια, ένα, μια υπηρεσία ανεξάρτητη. Καλά, καλά. Προτείνεται λοιπόν μια προφορική τροποποίηση για την παράγραφο 6. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Θα την ψηφίσουμε μετά τις τροπολογίες. Λοιπόν, αρχίζουμε με την τροπολογία 1 του κυρίου Γκέγερ. Avec l'amendement oral de, du rapporteur. Qui est pour Υπέρ. Κατά. Ποιες εγκρίνεται. Μετά τρεις τροπολογίες της κυρίας Τράουτμαν μπορούμε μαζί. Όχι. Ο, καλά, καλά. Τροπολογία 2. Υπέρ. Η εσύ είναι κατά. Κανείς, απολύτως κανείς καημένη Κατερίνα. Λοιπόν, τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Α, α, α, επαλήθευση. Τροπολογία 3. Τροπολογία 3, ε. 3. Ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά. Μάλιστα. 10 υπέρ, 11 κατά. Η αριστερά έχει καταψηφίσει την κυρία Τράουτμαν. Τέσσερα η είναι επίσης κατά. Κανείς πάλι. Κανείς. Κανείς. Κατά. Ε, αποχές. Εντάξει. Αποχές. Προφορική τροποποίηση τώρα της Γιούτα Χάουγκ που προσθέτει στην παράγραφο 6 για να μετατραπεί τον Μπερέκ σε ένα σώμα με πραγματικές δικαιοδοσίες ανεξάρτητο των ευρωπαϊκών θεσμών και κρατών. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ποχέ. Μία ψήφη κατά, μία αποχή εγκρίνεται. Να το δακτυλογραφήσετε δεόντως λοιπόν, ωραία. Συγχαρητήρια στην Χιούτα. Α, όχι και τελική ψηφοφορία, τελική, τελική. Τελική και ηλεκτρονική για την ομοδότηση της Χιούτα Χάουγκ. Εκεί. Λοιπόν, 20 ψήφοι υπέρ, ουδεμία κατά μία αποχή. Τρίαμβος. Κάρα Λοιπόν, έχουμε και άλλη μια ψηφοφορία που σας προτείνω σε συμφωνία με τους συντονιστάς. Είναι για το σημείο 9. Η γδομοδότησή μας δηλαδή για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για μια χρηματοδοτική ενίσχυση σε τρία, για τρία κράτη-μέλη. είναι βασικά το νομική, η νομική πτυχή του συμπληρωματικού 7. Σας υπενθυμίζω ότι ο συμπληρωματικός και περιοριστικός πληγισμός 7 είναι τμήμα του Ποδούπου. Εμείς θα ψηφίσουμε στις 5 Νοεμβρίου, στις 5 Νοεμβρίου το απόγευμα και στην Ολομέλεια 19 Νοεμβρίου. Αλλά και όμως έχουμε μια γνωμοδότηση να εγκρίνουμε για το νομικό υπόβαθρο προς την Επιτροπή Περίφ και πρέπει να την εγκρίνουμε έγκαιρα ώστε η Περίφ να μπορέσει να ψηφίσει έγκαιρα και εκείνη και τα προγράμματα του διορθωτικού ΕΠΤΑ να εφαρμοστούν εγκαίρως και αυτά. Είναι συντάκτης ο Ράιμερ Μπέγκερ, τον, Μπέγκερ τον οποίο αντικαθιστά η συθονία. Χωρίς τροπολογίες. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαίρουμε λοιπόν και τη Σιδονία και όλους. Λοιπόν. Το 23 και 24 τώρα που είναι μεταφορές ε, πιστώσεων. και 24. Τζοβάνι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχουμε δύο αιτήσει επιστροφών 22 μετά από επίσημο αίτημα της, ε, ε της, της, ε, μία μεταφορά όσον αφορά την βοήθεια στην ε, ανάπτυξη της υπαίθρου και που θα πηγαίνει στην ε, μία μεταφορά λοιπόν για τα κοινωνικά ταμεία θα σχετίζεται με συγκεκριμένα προγράμματα, μικρό ρυθμό προγραμμάτων υποδομής στην δημοκρατία αυτή την ΦΥΡΟΜ παρόμοια με προηγούμενα προγράμματα. Πρόκειται για 18 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ προτείνω να υπερψηφίσουμε αυτή τη μεταφορά. Να σας παρουσιάσω και το επόμενο αίτημα μεταφοράς. Ναι, το ένα αφορά ε, την, την μεταφορά υπαριθμών 27 που αφορά την ε, Κομμονίτα Βαλενθιάνα. 840 εκατομμύρια ε, που θα καλύψει ένα συντονισμένο πακέτο ε, προσωπικών υπηρεσιών ε, που αφορούν απολυμένους από 140 επιχειρήσεις ε, που προέρχονται από μη μεταλούχα υλικά εξόριξης. Πρόκειται για απολυμένους λοιπόν που θα τους βοηθήσουν τα προγράμματα αυτά να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας. Αυτό το δεύτερο, αυτή η δεύτερη μεταφορά είναι η παριθμόν 27, αλλά να ξεκινήσουμε από τη μεταφορά η παριθμόν 22 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Μεταφορά η παριθμόν 27 υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται ε, ίδια ψηφοφορία με την προηγούμενη έκθεση ε, Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε Τζοβάνι. Ε, Χάιντερ θα μας παρουσιάσεις ε, όλες τις μεταφορές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ναι, είναι δύο οι μεταφορές αυτές των 5.000 και 45 συν 56 είναι διπλή και η Επιτροπή Περιφερειών που ζητάει 75.016, 94 και τα λοιπά και 50 κάτι. Ε, είναι μικρές μεταφορές. Συμφωνεί ο εισηγητής που δυστυχώς απουσιάζει γιατί κολλείεται. Δεν χρειάζεται περισσότερες λεπτομέρειες. Τις έχω άμα θέλετε, αλλά όλοι ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Ε, je vous propose de voter... Τώρα σας προτείνω να ψηφίσουμε ανα, ή, ανα όργανο. Λοιπόν, ψηφίζουμε τις δύο μεταφορές 5 και 6 του δικαστηρίου. Υπέ, Κατά. Ποιες εγκρίνονται. Μετά οι μεταφορές 9, 1, 2 και 3. Οι μεταφορές INF. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Πάνε και αυτά. Ευχαριστούμε Χάιντερ. Τελείωσαν λοιπόν οι ψηφοφορίες και τώρα περνάμε στο σημείο 10, δύο εκθέσεις της κυρίας Καρβάλιο. Πρώτα για το πρόγραμμα Κοπέρνικος. Ο Κοπέρνικος έχει διαδεχθεί το προηγούμενο πρόγραμμα GMPS. Είναι πολύ χρήσιμο πρόγραμμα που δίνει πληροφορίες και δεδομένα από παρατήρηση από το διάστημα αλλά και για προστασία του περιβάλλοντος, αντιμετώπιση των κλιματολογικών αλλαγών, έλεγχο της κυκλοφορίας, πολλές εφαρμογές του μπορούν να γίνουν. Και έχει όντως συνεισφέρει σε οικονομική ανάπτυξη πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα. Είναι πολύ σημαντικό πρόγραμμα διαστημικό. Έχει δική του γραμμή στον προϋπολογισμό με ποσόν 3,786 εκατομμύρια είχε το 11, σε τιμές του 11 ή 4,921 τώρα. Η τωρινή πρόταση της Κομισιόν κατατέθηκε μετά από τη λήξη των διαπραγματεύσεων με το, για το Και το ποσό είναι καθορισμένο. Στη γνωμοδότησή μου λοιπόν τονίζω τρία πράγματα. Πρώτον, την θέση της έκθεσης Πολδίπ. Ενώ ταυτόχρονα ζητούμε να μην μειωθούν άλλα προγράμματα όπως της έρευνας λόγω της ανάπτυξης του Κοπερνίκου. Επομένως, τα διαθέσιμα περιθώρια θα έπρεπε κανονικά να αρκέσουν. Δεύτερον, είναι σημαντικό να αποφύγουμε πρόσθετο κόστος για να είναι πιο εύκολος ο έλεγχος και γι' αυτό κατανέμονται σε διάφορες κατηγορίες οι δραστηριότητε του Κοπερνίκου. Και τρίτον και τελευταίον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να παίξει σημαντικότερο ρόλο στην επιτήρηση, εποπτεία και έλεγχο της ανάπτυξη του προγράμματος. Η Κομισιόν πρέπει εγκαίρω να μα δώσει όλες τι απαραίτητε πληροφορίε για το πρόγραμμα ιδιαίτερα τη διατήρηση κινδύνου, κόστος, ραγματισμό κλπ. Αυτά έβαλα στην ομοδότησή μου. Σας κατευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ κύριε εισηγήτρια. Ο κύριος Μινά ζήτησε το λόγο. Μα ευχαριστώ πρόεδρε κυρίες και κύριοι. Επιτρέψτε μου λίγο να συμπληρώσω. Ένα σημαντικό στοιχείο για την ασφάλεια του προγράμματος. Είναι πολύ σημαντικό να είναι αυτή δεδομένη. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε και να αξιοποιήσουμε την εμπειρία και την υποδομή που έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια του προγράμματος Έγνος και Γαλιλαίο, που είναι αντίστοιχα με το Ποκοπέρνικο. Όταν ε, μελέτησα αυτό το θέμα, προσέκουσα ρούσας ε, έλλειψη κατανόησης από το κοινό για αυτά τα προγράμματα. Και αυτό τι σημαίνει. Ε, με επιβεβαίωσε στην άποψη που είχα ότι πρέπει να ενημερώνουμε καλύτερα τον κόσμο για το ρόλο των προγραμμάτων και των προϊόντων που έχουν να κάνουν με το διάστημα και πώς επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή. Θα πρέπει να υπερασπιζόμαστε τα κονδύλια που ε, δαπανούμε για αυτά τα προγράμματα και να το εξηγούμε στον κόσμο. Θα πρέπει να επιφορτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτό το έργο, αυτή την αποστολή. Και θα παρακαλούσα να ενημερώνουμε καλύτερα και να συμπεριλαμβάνεται και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος. Προς την κατεύθυνση αυτή λοιπόν έχω ήδη καταθέσει τροπολογία που στοχεύει στην ενημέρωση ακριβώς του Κοινοβουλίου ε, με ε, βάση τους ελέγχους που κάνει το ελεγκτικό συνέδριο και η Όλαφ. Αυτά τα ελέγχει η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, έτσι καλώ στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την καλή της πραγματογνωμοσύνη και την καλή συνεργασία που είχαμε ε, μεταξύ μας. Ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Η κυρία Καρβάλιο σημείωσε τις προτάσεις σας. Οπότε, για το θέμα αυτό, για το θέμα αυτό βεβαίως, βεβαίως, δεν θα ψηφίσουμε. Προθεσμία κατάσταση τροπολογιών. Α, συγγνώμη. Η Αν Γένσεν είχε ζητήσει το λόγο αν είναι δυνατόν. Πώς δεν σε είδα. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτά ε, που ακούστηκαν για τις διαστημικές πολιτικές και πόσο σημαντικό είναι. Έχω μια ερώτηση όμως για την κυρία Καρβάλιο, διότι είναι γεγονός ότι ε, υπήρχε ο Γαλιλαίος, αυτό το πρόγραμμα το GMES ε, και κάπου είναι ίδια τα χαρακτηριστικά τους. Όταν μιλούμε για υπέρβαση ε, κονδυλίων, τι εννοούμε, έχω την αίσθηση ότι αυτό το πρόγραμμα συνενώνει πολλά μικρά έργα και δεν έχουμε δει στο παρελθόν να υπερβαίνει το κόστος. Και θα ήθελα κάπως να μας διαβεβαιώσουν ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό και στο μέλλον. Να υπάρχει ε, μια ευελιξία στον τρόπο που στείνεται το πρόγραμμα για να προσαρμόζεται καλύτερα στο κόστος. Δεν είναι σαν τον Γαλιλαίο που ε, μας ζητούν ε, συνέχεια λεφτά, διότι αλλιώς θα χαθούν αυτά που ήδη έχουν δαπανηθεί μέχρι τώρα. Θα πρέπει να είμαστε έτσι προσεκτικοί σε αυτό. Χωρίς να μας τρομοκρατεί η υπέρβαση του κόστους. Γιατί δεν την έχουμε δει μέχρι τώρα και κάπως υπάρχουν και εγγύσεις ότι δεν πρόκειται να τη δούμε και στο μέλλον. Κυρία Καρβάγιο, θέλετε να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, καλοδεχούμενες οι προτάσεις του σκιώδου συγητού. Όσο γίνεται να χρησιμοποιήσουμε την ίδια υποδομή του Γαλιλαίου και να ενημερώνουμε καλύτερα τον κόσμο και την Επιτροπή Ελέγχου για τον έλεγχο που διεξάγει Όλαφ. Ήδη υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας που μπορούν να αξιοποιηθούν και να ενισχυθούν να χρειάζεται. Συμφωνώ απολύτως με το ζήτημα που λέγει ότι δεν υπάρχει ο ίδιος κίνδυνος ε, υπέρβασης του κόστους όπως ο Γαλιλαίο ή είναι πιο μικρής κλίμακας ε, έργα αυτά και σε όλα τα project έχουμε κάποιες τροπολογίες που να μας βεβαιώνουν ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση κόστους και δεν θα Αντληθούν κονδύλια από άλλα έργα που είναι πάρα πολύ σημαντικά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως είναι ε, Ορίζον 2020 και τα σχετικά έργα. Είναι πολύ μικρότερος ο κίνδυνος από ό,τι με το Γαλιλαίο έτσι κι αλλιώς πάντως. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ναι. ε, ανακεφαλαίωσης. Θυμίζω ότι το χρονοδιάγραμμα για την έκθεση Καρβάη έχει ως εξής προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 24 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Θα ψηφίσουμε στις 14, είναι στο 14 Όχι στις 5, στις 14 Νοεμβρίου, ήτρε ψηφίζει 28, η δε ολομέλεια ακόμα δεν έχει οριστεί. Σε ό,τι αφορά τώρα το σημείο 11 και άλλη έκθεση κυρίας Καρβάλιο είναι αυτή για την ε, παρακολούθηση του διαστήματος. Παρακαλώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και αυτή η έκθεση αφορά ένα σημαντικό ε, ζήτημα. Ένα πρόγραμμα το οποίο θέλει ε, να συμβάλλει ε, στην οικοδόμηση μιας ανεξάρτητης ευρωπαϊκής ικανότητας επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος που θα αποσκοπεί κυρίως στην αποτροπή συγκρούσεων στο διάστημα. Uh, ε, βασιζόμαστε σε έκθεση της Ευρωπαϊκής ε, πρόταση συγγνώμη, της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής που αποσκοπεί στην, στην δικτύωση κατά κάποιο τρόπο των υφισταμένων δομών και που προτίθεται να δώσει περίπου 70 εκατομμύρια σε μια επταετή περίοδο. Δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσό αν αναλογιστούμε τους στόχους που έχουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε παρακολούθηση του διαστήματος, να επιτηρούμε τους κινδύνους ε, σύγκρουσης ε, πρόκειται για διαστημικό εντό εισαγωγικών ε, πρόγραμμα. Το ερώτημα εδώ είναι ότι ε, στη Draft Legal Act δεν υπάρχει ε, προϋπολογισμός. Ε, γι' αυτό εγώ υποβάλλω τροπολογία έτσι ώστε ακριβώς να αναφέρω τα 70 εκατομμύρια στην επταετή περίοδο ποσό το οποίο αναφέρεται στο επεξηγηματικό υπόμνημα της Κομισιόν. Αλλά θέλουμε να ξέρουμε από πού προέρχονται τα χρήματα αυτά. Θα υποβάλουμε λοιπόν και μια τροπολογία η οποία θα λέει ότι αυτή η χρηματοδότηση προέρχεται κυρίως από τον Γαλιλαίο και τον Κοπέρνικο γιατί είναι άμεσα συνδεδεμένα διαστημικά προγράμματα και ότι επίσης θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε όσον αφορά την έρευνα γιατί και εδώ υπάρχουν, υπάρχει ανάγκη έρευνας ε, στο, για το διάστημα ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν για τα ερευνητικά προγράμματα κονδύλια των τον ε, ορίζοντα 2020 ε, καθώς επίσης και από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Αλλά τα περισσότερα χρήματα θα έρθουν από τον Γαλιλαίο και τον Κοπέρνικο. Τρίτον, η Draft Legal Act ε, δεν αφορά την ε, ε, κατάτμιση του προϋπολογισμού αναδραστηριότητα και επομένως γι' αυτό ακριβώς ζητήσαμε μέσω τροπολογίας να αναφερθούν αυτά τα τρία τμήματα της έρευνας τα οποία θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικά και τα οποία θεωρούμε ότι θα δώσουν μεγαλύτερη διαφάνεια στην και λογιστική καθημερινότητα καθαρότητα στους, ε, στο λογαριασμό αυτό. Λοιπόν, εν συνόψη, θα έχουμε τα 70 εκατομμύρια ε, σε επταετή περίοδο. Θα ε, ζητήσουμε αποσαφηνήσεις για το από πού προέρχονται τα χρήματα αυτά και μία στόχευση όσον αφορά την δαπάνη των χρημάτων αυτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια ο κύριος Μινάρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να κάνω και εγώ κάποιες συμπληρωματικές παρατηρήσεις σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Καρβάλιο. Όπως και, στο προηγούμενο, και για το προηγούμενο σημείο χαίρομαι που έχουμε την πρόταση αυτή ε, και η οποία θα διευρύνει την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο διάστημα. Οι διαστημικές δραστηριότητες, δηλαδή δραστηριότητες σχετιζόμενες με το διάστημα είναι ε, ένα σημαντικό κεφάλαιο της οικονομικής ζωής και μπορούν να ε, βοηθήσουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που όλοι θέλουμε. Ε, θέλουμε να προστατέψουμε τους υφιστάμενους και μελλοντικούς ευρωπαϊκούς δορυφόρους και μάλιστα να τους προστατέψουμε με αποτελεσματικό τρόπο. Ε, θεωρούμε ότι, όπως είπε και η συγγύτρια θα πρέπει ε, να υπάρχει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και επίσης μπορούν να γίνουν εξοικονομήσεις ε, από τα κράτη, για τα κράτη-μέλη τα οποία ε, θα εκμεταλλευτούν το σύστημα. Έχω υποβάλει τρεις τροπολογίες ε, όσον αφορά το, το, τη γνωμοδότηση αυτή σε συμφωνία και με την εισηγήτριά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ λέει ο Πρόεδρος. Πολύ καλή συνεργασία. Αγαστή συνεργασία λοιπόν μεταξύ των ειδημόνων του διαστήματος και χαίρομαι πολύ γι' αυτό και η προηγούμενη έκθεση και ε, τούτη εδώ ε, έχουν ίδια προθεσμία κατάθεση τροπολογιών την 24η Οκτωβρίου. 14 ε, Νοεμβρίου η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας και ψηφοφορία στην Ήτρε 28 Νοεμβρίου. Ευχαριστούμε την κυρία Καρβάλιο. Για το σημείο 12 τώρα. Ο κύριος Σέντερντεν δεν είναι εδώ. Euh, Αλλά ο, ο συνέλφος ε, Κάλφιν τον ε, αντικαθιστά και θα μας ε, παρουσιάσει λοιπόν αυτήν την γνωμοδότηση, η ικανότητα των κρατών μελών της Ένωσης να αρχίσουν εν τη νέα περίοδο προγραμματισμού της πολιτικής για τη συνοχή και με την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα. Πολύ σημαντικά θέματα. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος του συναδέλφου μου Φρεντερίκ Νταρντέν θα σας περιγράψω τη γνωμοδότησή του. Διαβάζω τι μου είπε να διαβάσω. Λοιπόν, καλό θα ήταν να τονίσουμε στη γνωμοδότηση αυτή ορισμένες προτάσεις που να ανταποκρίνονται στις φημερινές δυσκολίες εφαρμογής της πολιτικής συνοχής στα κράτη-μέλη. Πρέπει να επιθυμίσουμε ότι στην πολιτική συμφωνία της 27 Ιουνίου για το ΣΕΦΠΕ ήδη εμφαίνονται τέτοιες προτεραιότητες για να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η νέα πολιτική συνοχής και τονίζουμε ότι αργά ή γρήγορα στον προϋπολογισμό θα γίνει μια συγκέντρωση των κονδυλίων. Είναι αναμφίβολο ότι στο τέλος της χρήσης 7-13 κατά δύο τρίτα τα κονδύλια αυτά αφορούν άμεσα την πολιτική συνοχή και πρέπει να αποφευθεί ο κίνδυνος μπλοκαρίσματος των προγραμμάτων της Ένωσης λόγω έλλειψης πληρωμών. Επίσης νομίζω ότι θα έπρεπε να βελτιωθεί η διαχείριση των τοπικών και περιφερειακών αρχών ήδη και η συμβολή τους ήδη από την περιγραφή, την υποβολή των προγραμμάτων μέχρι και την εφαρμογή τους για να υπάρξει καλύτερη διαχείριση της νέας πολιτικής συνοχής αυτή η αυξημένη αποτελεσματικότητα των επενδύσεων της Ένωσης θα ενδυναμωθεί και από τη μεγαλύτερη συνέργεια μεταξύ του ενωσιακού προπολογισμού και των προϋπολογισμών των χωρών μελών και των ε, τοπικών και αρχών. Η Κομισιόν πρέπει εδώ να μας δείξει, με ποιον, το μας πει ποιον τρόπο θα ενδυναμωθεί η χρήση και η λειτουργία του ενωσιακού προϋπολογισμού για να μην δε αποθαρρυνθούν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές σας υπενθυμίζω ότι υπάρχει και η αρχή της αιρεσιμότητας. Επίσης πρέπει να τονίσω ότι είναι απαραίτητο και η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να απλοποιήσουν τις διαδικασίες και τους κανόνες για τις δημόσιες προμήθειες ή αγορές καθώς και τους υποπτικούς μηχανισμούς. Αυτά μου είπε ο Φρεντερικ να διαβάσω, αυτά διάβασα. Ναι. Και ζητάει συγγνώμη που δεν μπόρεσε να προσέλθει γιατί είναι στη Λιέχη με τον πρόεδρο Βαρόσο. Ευχαριστώ. Κατανοητό. είχε και την ευγένεια να μας ενημερώσει προηγουμένως. Ευχαριστώ Βάιλο για αυτή την παρουσίαση. Δεν ζητεί κανείς το λόγο. Θαυμάσια. Α, ζητάει. Ε, να κοίταζα και όλες ο κύριος Κοσλόφσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Νταρτέν ε, έθεσε πολύ σωστά κάποια ερωτήματα και κάποια ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη από την Περιφερειακή Επιτροπή όταν θα κληθεί να ψηφίσει. Συμφωνώ πολύτως με την έμφαση που δίδεται στη λεγόμενη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην πολιτική συνοχής ε, επίσης συμφωνώ ότι οι αρχές τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης θα πρέπει πλήρως να συμμετέχουν στα επιχειρησιακά προγράμματα από την αρχή μέχρι το τέλος τους σε όλες τις φάσεις και ε, στην αξιολόγηση εκ των υστέρων. Θα πρέπει να δίδεται όσο γίνεται μεγαλύτερη υποστήριξη ε, στις ΟΤΑ και στις περιφερειακές αρχές για να μπορούν να συγχρηματοδοτούν ε, τα μεγάλα μικρότερα έργα. Η οικονομική διαχείριση δεν θα πρέπει να έχει αρνητικές επιπτώσεις ε, στα οικονομικά των ε, δήμων και των περιφερειών. Σε ό,τι αφορά το αποθεματικό επιδόσεων, ε, όπως πρότεινε η πολωνική κυβέρνηση, θα πρέπει να αποτελεί αυτή ένα χέγγιο για τους δικαιούχους και το μέσον αυτό, εάν δημιουργηθεί σωστά, θα βελτιώσει τη χρήση και τη διαχείριση των διασωτικών πόρων. Πολύ ωραία. Άψογα. Λοιπόν, για την έκθεση αυτή του κ. Νταρντέν, ορμοδότης. Είναι παρόμοιο το χρονοδιάγραμμα με της κυρίας Καρβάλιο. 24 Οκτωβρίου στις 6 λίγη διόρια κατάσταση τροπολογιών, 14 Νοεμβρίου στην Επιτροπή Πολιτισμών, η οποία θα και στην Περιφερειακή 28 Νοεμβρίου, ολομέλεια δεν έχει ακόμη καθορίστη. Ευχαριστούμε Ιβαϊλό τελευταίο σημείο, το 14, όχι το 13 και 14, δύο πρωτόκολλα για την αλληλεία με το Γαβόν και με το Βασίλειο του Μαρόκου. Ο κύριος Αλφόνση είναι εισηγητής και για τη Δημοκρατία και για το Βασίλειο, αλλά η Ισαβέλα Δουράν θα τον αντικαταστήσει. <laughs> του βασιλείου του Βελγίου. Λοιπόν, αντικαθιστώ εδώ τον κύριο Αλφόνση που κολλείεται. Για το πρωτόκολλο με το Γαβόν πρόκειται για ανανέωση ενός προηγούμενου πρωτοκόλλου αλίας μεταξύ Ένωσης και Γαβών που αφορά τρία χρόνια και προβλέπει μία αποζημίωση 4,1 εκατομμυρίων προς το γαβόν για να επιτρέπεται στα ευρωπαϊκά αλλιευτικά πλοιάρη να αλλιεύουν στα χωρικά ύδατα του γαβόν σύμφωνα με τα κριτήρια της βιωσιμότητας. Ο εισηγητής λοιπόν, ο κ. Αλφόνση δηλαδή, ζητάει από την Κομισιόν να επιτηρεί την εφαρμογή της συμφωνίας του πρωτοκόλου μάλλον και να βλέπει αν όντως γίνονται σεβαστές οι ρήτρες για τα ευρωπαϊκά πλοιάρια και να κάνει ανάλυση και αξιολόγηση κόστους ωφέλους. Συστήνουμε λοιπόν η Επιτροπή μας να εγκρίνει το πρωτόκολλο αυτό. Και η διορία κατάσταση είναι λύγει 28 Οκτωβρίου. 22. 22. 22. Α, μάλιστα αυτά για το Γαβόν. Να συνεχίσω με το Μαρόκο. Α, λοιπόν. Και εδώ είναι ένα πρωτόκολλο που ακολουθεί την αποτυχία του προηγουμένου πρωτοκόλλου. Γιατί είχε αρνηθεί το Μαρόκο διότι είχε γίνει μια αρνητική αξιολόγηση κόστου ωφέλους, είχε αμφιβολίες στο κοινοβούλιο ως προς τους αλλιευτικούς πόρους και δεν είχε ληφθεί καθόλου υπόψη το πρόβλημα της δυτικής Σαχάρας. Η Επιτροπή λοιπόν η Κομισιόν θέλει σε νέα, να δώσει μια νέα μορφή σε αυτό το πρωτόκολλο τη μείωση του αριθμού των ευρωπαϊκών πληρών που θα έχουν το δικαίωμα να αλλιεύουν στα χωρικά ύδατα τα δυτική Αγάρας και του Μαρόκου και όλες οι αντιρρήσεις του Κοινοβουλίου αλλά όλες οι αντιρρήσεις του Κοινοβουλίου δυστυχώς δεν έχουν απαντηθεί η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου είχε καταλήξει ότι πρέπει να υπάρξει συμφωνία με τη Δυτική Σαχάρα και να τύχει και διαβούλευση. Ενώ οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν έχουν καν δεχτεί να λάβουν υπόψη τους την περιφέρεια αυτή. Η αξιολόγηση κόστους ωφέλους ανεξάρτητα έγινε ανεξάρτητα και σε χωρίς σχέση με το πρώτο προηγούμενο πρωτόκολλο και κατέληξε ότι είναι αρνητική Ανετικό το συμπέρασμα. Στο νέο πρωτόκολλο δεν φαίνεται γιατί άλλαξαν τα πράγματα. Γιατί. Ο εισηγητής δεν βρήκε στοιχεία που να δείχνουν ότι υπάρχει καμία βελτίωση ενώ πρόκειται για 120 εκατομμύρια ευρώ εδώ πέρα. Τέλος, ένα θέμα που ίσως δεν είναι και τόσο θέμα δικό μας είναι υπεραλίευση. Αυτό είχαμε πει ότι θέλαμε να ληφθεί υπόψη γιατί ορισμένα αποθέματα ηχθείων μπορεί να τη χάνουν υπερβολικής εκμετάλλευσης. Ο εισηγητής δεν έμαθε τίποτα καινούριο τα τελευταία αυτά χρόνια για την κατάσταση των αποθεμάτων στα χωρικά του Μαρόκου και της Δικής Σαχάρας και για αυτούς τους λόγους ο κύριος Αλφόνση ζητά απόρριψη και 22 Οκτωβρίου λίγη διορία κατάθεση τροπαλογιών. Πρόεδρος Άψογα. Λοιπόν, συνοψίζω. Ο εισηγητής προτείνει θετική απόφαση για το Γαμπόν και αρνητική για το Μαρόκο. Θέλει κανείς το λόγο? Όχι. Όπως είπε η κυρία Τουιρόν, προθεσμίες 22 Οκτωβρίου το μεσημέρι και για τις δύο εκθέσεις για τις τροφολογίε. ψηφοφορία στην Επιτροπή Προπολογισμού στις 14 Νοεμβρίου εν ώψη ε, ψηφοφορίας από τη ουσίας στην Επιτροπή στι 27 Νοεμβρίου. Πολύ ωραία, νομίζω ότι έχουμε εξαντλήσει την ημερήσια διάταξη. Σας ευχαριστώ. Λήξη στις συνεδρίες.